So, wir können wieder starten, Λοιπόν, α ξαναρχίσουμε συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι. Δεν θέλω να καθυστερήσουμε πολύ. Έχουμε την έκθεση στην ημερήσια διάταξη που είχαμε αναβάλει. Να σας πω ποια έκθεση είναι. Διευρωπαϊκό Δίκτυο Τηλεπικοινωνιών και κατάργηση της απόφασης υπαριθμών ΤΑΔΕ 133697. Εισηγητή είναι ο Ρέστε Ρώση και θα ήθελα να του δώσω μέσα στο λόγο. Παρακαλώ, κύριε Ρώση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αυτό το σχέδιο γνωμοδότησης αφορά τα Ευρωπαϊκό Δίκτυο Τηλεπικοινωνιών και την κατάργηση της απόφασης 1336 το 97. Θα έλεγα καταρχάς πως το κείμενο είναι καλογραμμένο, τονίζει την ε, ανάγκη παροχής ε, ίντερνετ σε όλους ε, την, για τη διάδοση των ευρωζωνικών δικτύων για να υπάρχουν υπηρεσίε ηλεκτρονικής δημόσιας διοίκησης και να βοηθηθεί επίσης και η υγειονομική βοήθεια μέσω διαδικτύου. Το είχαμε θίξει το ζήτημα όταν εξετάσαμε το θέμα των ατόμων με αναπηρία. Θα ήταν χρήσιμο λοιπόν να να διασυνδέονται με κοινά δίκτυα ώστε σε πραγματικό χρόνο να έχουν οι γιατροί και τις προφορίες ε, για τους ασθενείς θα μπορούν ε, με αυτόν τον τρόπο οι πολίτες να επιλέγουν την χώρα στην οποία θέλουν ε, να νοσηλευτούν ή να θεραπευτούν. Οι τροπολογίες ε, πηγαίνουν προς την κατεύθυνση αυτή, αλλά ζητούν επίσης να αποδοθεί ιδιαίτερη προσοχή από πλευράς κομισιών για το πώς θα πρέπει να αντιμετωπίζουν τα δεδομένα που θα αποστέλλονται. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει μια μιογενής παρουσίαση επειδή πρόκειται για δεδομένα ευαίσθητα και ενδεχόμενα, επιδεχόμενα μάλλον ποικίλων ερμηνεών θα πρέπει λοιπόν να έχουν την κατάλληλη μορφή. Θα υπάρχει και, και μια κωδικοποίηση κοινή έτσι ώστε να υπάρχει ένας ενίος και τρόπος για την ανάγνωση αυτών των εγγράφων τα οποία θα αποτελούν το βασικό προφίλ του ασθενούς που περιλαμβάνει διαλειτουργικές και υπηρεσίε, υπηρεσίες, για παράδειγμα αιματολογικοί παράγοντες, ιστορικό κλπ. Ζητάμε λοιπόν να υπάρξει ένας κωδικός ευρωπαϊκός μόνο σήμαντος που θα μπορούν οι Ευρωπαίοι πολίτες να τον μεταχειρίζονται να τον χρησιμοποιούν μάλλον και με τις επαφές που θα έχουν με τις ε, επιμέρους διοικήσεις. Ένα άλλο ζήτημα το οποίο κρίνω ότι είναι εξίσου σημαντικό συνδέεται με το ότι δεν ε, θα πρέπει να αναθέτουμε στην Κομισιόν την εξουσία για έκδοση πράξεων κατεξιοδότηση για τροποποίηση του περιεχομένου του παραρτήματος. Νομίζουμε ότι θα είναι καταλληλότερο γι' αυτό το λόγο η συνήθι νομοθετική διαδικασία. Οι τροπολογίες λοιπόν που έχω καταθέσει ε, βαίνουν ακριβώς προς αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή να καταργηθούν ε, οι πράξεις κατεξιοδότηση που δύναται να εκδίδει η Κομισιόν. Παναλαμβάνω ότι εγώ τονίζω το, θέμα των ε, πράξεων κατεξοδότηση και των ε, κοινών κανόνων που θα πρέπει να διέπουν την ε, ανταλλαγή αυτών των, την υποβολή με αυτών των δεδομένων άμεσα στα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ τον ε, εισηγητή και πάμε τώρα στους σκιώδεις εισηγητές. Ε, συνάδελφος Αντωνέσκου για το ΕΛΚ, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πράγματι, το οικονομικό αυτό μέσω της Επιτροπής ε, μπορεί να λύσει ε, τα προβλήματα που δημιουργούνται από την απουσία μιας ισχυρής υποδομής. Ε, υπάρχει έλλειψη ανταγωνισμού, σημαντικός κίνδυνος ε, στην αγορά και οι ε, κοινοφιλείς επιχειρήσεις δεν είναι αρκετά ανεπτυγμένες λόγω του κατακαιρματισμού των τεχνολογικών λύσεων. Η χρήση διαρθρωτικών ταμείων για την υποδομή στις ψηφιακές υπηρεσίες δεν μπόρεσαν να ε, οδηγήσουν στην κρίσιμη μάζα που θα ήταν απαραίτητη για την ε, σωστή διάδοση των ε, ψηφιακών υπηρεσιών. 9,2 εκατομμύρια έχουν προβλεφθεί ενώ οι πραγματικές ανάγκες είναι 270 εκατομμύριων ευρώ και γι' αυτό πιστεύουμε ότι ο μηχανισμός αυτός θα πρέπει να θεωρηθεί συμπληρωματικός ώστε να ευαισθητοποιήσει το κοινό απέναντι στην ανάγκη για περαιτέρω επενδύσεις. Ιδιαίτερα ε, στις πέτρες περιοχές υπάρχει ε, μεγάλη ανάγκη. Όσον αφορά την τροπολογία, την, ε, συγγνώμη, την υποδομή θα πρέπει η το πρόβλημα είναι ότι οι ιδιώτες επενδυτές δεν επενδύουν λόγω του ότι οι επενδύσεις αυτές δεν συμφέρουν πολύ. Θα πρέπει να έχουμε μια μη διακριτική πολιτική για να μειώσουμε το χάσμα ανάμεσα στους ε, ιστορικούς φορείς και τους ε, ανταγωνιστές τους, ιδιαίτερα όσον αφορά τα δίκτυα, ε, τα για το διαδίκτυο. Τα ε, προγράμματα που θα εφαρμοστούν θα πρέπει ε, τεχνολογικά να είναι ουδέτερα και χρειαζόμαστε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των ε, νέων αυτών μέσων καθώς και τη δύναμη μόχλεσής τους, διότι χρειαζόμαστε συντονισμό των ταμείων που προβλέπει ο κανονισμός αυτός και των πόρων που προβλέπουν άλλες πρωτοβουλίες για να αποφύγουμε ε, την επικάλυψη εργασιών ε, ή ε, το να ξεχαστούν κάποιες συγκεκριμένες περιοχές, κάποιοι, κάποιοι Σημαντικό είναι να μπορούν να χρησιμοποιηθούν και, και πόρια από τα διαφροντικά ταμεία και από το Ταμείο Συνοχής. Όσον αφορά τα προγράμματα κοινή ωφελία στον τομέα των ψηφιακών υπηρεσιών, θα πρέπει να συμπεριληφθούν εδώ και διάφορες υπηρεσίες όπως είναι η ηλεκτρονική υγεία. Και θα ήθελα να επικροτήσω τις τροπολογίες 12, 13 και 14, διότι γνωρίζουμε ότι οι εφαρμογές υγείας ε, παίζουν όλο και πιο σημαντικό ρόλο στην, ε, στη γιατρική. Θέλουμε περισσότερε πληροφορίε από την Κομισιόν σχετικά με τα κριτήρια που προβλέπουν ε, για να καθοριστούν ε, οι τομεί αυτού ιδιαίτερου ενδιαφέροντος. Ε, και με ενδιαφέρει επίση να ακούσω γιατί η Κομισιόν δεν έχει προβλέψει ένα πρόγραμμα που να λέγεται ηλεκτρονικό περιβάλλον, όπω έχουμε αυτό για την ηλεκτρονική υγεία. Όσον αφορά τις αρμοδιότητες επιτροπής σε σχέση με τον κανονισμό αυτό, και σύμφωνα με την πρόταση, είναι πολύ ευρείες οι αρμοδιότητες αυτέ. και ο η επιλογή των προγραμμάτων εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Κομισιόν. Είναι ένας ε, τομέας ε, πολύ δυναμικός ε, που αναπτύσσεται ραγδαία. Γνωρίζουμε την ανάγκη να έχουμε ένα ευέλικτο μέσο Χρειαζόμαστε όμως επίσης και νομική βεβαιότητα, καθώς και προβλεψιμότητα για τις επενδύσεις και γι' αυτό θα πρέπει να σκεφτούμε πολύ προσεκτικά τον μηχανισμό για τον έλεγχο των αρμοδιοτήτων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε η κυρία Πόσπαχ, ο κύριος Πρόντι. Όχι, γιατί για... τότε η, η Λίντα Μακάβαν εκπροσωπεί τον Βιτόριο Πρόντι. Ευχαριστώ. Κολλείεται ο κύριος Πρόντι δυστυχώς ε, σήμερα και μου ζήτησε να πω τα εξής στους συναδέλφους της Επιτροπής πιστεύουμε ότι ε, τα ευρωζωνικά δίκτυα θα είναι προς όφελος μείωσης του κόστους ε, των ε, υπηρεσιών και θα ξεπεράσουμε έτσι το ψηφιακό χάσμα στην Ευρώπη, ιδιαίτερα στην Ήπεθρο. Το παράρτημα στην Πρώτη Ευρωπαϊκή Επιτροπή τονίζει ότι οι υπηρεσίες ευρυζωνικότητας θα βελτιώσουν τη ζωή των πολιτών. Ωστόσο, έχω κάποιες ανησυχίες για τα όσα λέει το παράρτημα. Ιδιαίτερα επειδή γίνεται η διαφοροποίηση και η ιεράρχηση προτεραιοτήτων είναι οριζόντιες οι προτεραιότητες γενικά για τις ψηφιακές υπηρεσίες και για την ευρυζωνικότητα. Αλλά δεν λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ποια είναι τα πιο σημαντικά και επίγοντα να γίνουν και ε, ποια θα πρέπει να γίνουν πρώτα. Αν δούμε τις άλλες πολιτικές στην Ένωση, όπω η ανακοινώσει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Περιφερειακή Πολιτική, την ψηφιακή ατζέντα για την Ευρώπη, τον οριζόντα για το 2020 και του στόχου του. Μπορούμε να αρχίσουμε με βάση τη σημασία του αυτά τα στοιχεία. Έχουμε και εμβληματικέ πρωτοβουλίε, όπω το GMES ε, και τέτοια αντίστοιχα, αλλά φοβούμε ότι αν επικρατήσουν αυτά, ε, τα θέματα που αφορούν την κοινωνία και την ενδιαφέρον περισσότερο θα χαθούν και θα μείνουν πίσω. Θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα σε βασικά έργα υποδομών για τα μικρά δίκτυα για τις, ε, την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και το μετριασμό των ε, συνεπειών σε όλες τις περιφέρειες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, θα πρέπει να έχουμε γρήγορο διαδικτύο για όλους, έρευνα ε, στις ε, τεχνολογίες, πληροφόρησης και επικοινωνίες και μια κοινωνία με λιγότερες εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Ο κύριος Ρώση, γιατί περιορίζεται μόνο στα θέματα της ηλεκτρονικής υγείας άραγε? υπάρχουν και άλλα στοιχεία που μπορούν να βοηθήσουν σε μια συστημική δυναμική κοινωνία όπως είναι η διάδοση ε, της γνώσης σε μια κοινωνία που βασίζεται ακριβώς σε αυτή. Χρειάζεται γενικότερη προσέγγιση, συνολικότερη. Είναι πολλά τα χρήματα που ε, δίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε αυτά τα σχέδια Αλλά όχι υπερβολικά λέει και ως πρώτη, γιατί είναι και οι στόχοι φιλόδοξοι. Δωρεάν roaming, ας πούμε, περιαγωγή στην κινητή τηλεφωνία. Ενώ ταυτόχρονα δίνουμε πολλά χρήματα σε ένα τομέα που έχει πολύ μεγάλο ορίζοντα μπροστά του. Τέλος, πώς μπορούμε να βεβαιωθούμε ότι οι βέλτιστες πρακτικές ακολουθούνται. Πώς μπορούμε να βεβαιωθούμε ότι δεν θα δαπανίσουμε 9,2 δισεκατομμύρια ευρώ και τελικά να ξυπνήσουμε την άλλη μέρα και να έχει ε, ε, ξεπεραστεί η τεχνολογία αυτή που θα έχουμε οικοδομήσει. Σε αυτούς τους τομείς που είναι τόσο ε, ραγδαία η εξέλιξη θα πρέπει να προσέχουμε που δίνουμε χρήματα. Το ξέρω, το έχω ζήσει στο πετσί μου. Το δημόσιο κάνει πολύ καιρό να πάρει μια ε, απόφαση για την επένδυση και μέχρι να γίνει αυτό ο ιδιωτικός τομέας έχει ξεφύγει, οι εξελίξεις τρέχουν και έχει ξεπεραστεί πλέον αυτή η επένδυση. Αυτά τα θέματα των μητρών ασθενών δεν ξέρω κύριε Ρώση, χρειάζονται προσοχή για τεράστια ηλεκτρονικά θέματα και προσπάθησαν στη χώρα μου να ψηφιοποιήσουν σε εθνικό επίπεδο του ε, τους φακέλους των ασθενών ήταν μια πανάκριβη προσπάθεια και τελικά μια τρύπα στο νερό. You know, ε, θα πρέπει να υποφελούνται οι πολίτες και από τις ιατρικές υπηρεσίες, οπότε δεν θα πρέπει να ε, δαπανούμε δισεκατομμύρια για να ψηφιοποιήσουμε όλες αυτές τις προφορίες για ορισμένους και μόνο. Δεν είναι καλύτερη χρήση των χρημάτων των φορολογουμένων σε αυτούς τους χαλεπούς καιρούς. Ξέρω ότι είναι μεγάλο το λόμπι, τα θυμάμαι πολύ καλά από την οδηγία για τις διασυνοριακές υπηρεσίες υγείας, αλλά πρέπει να προσέξουμε. Ευχαριστώ. Ρόσπαχ από την ομάδα της. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ε, μιλώ εκ μέρους ε, συναδέλφου που δεν μπορεί να παραστεί στη σημερινή συνεδρίαση της κυρίας Γιανακουδάκη. Όσον αφορά την ε, πρόταση της Κομισιόν, ε, θεωρείται σημαντικό βήμα ε, προς μια έννοια αγορά. Η πρόταση αυτή μπορεί να βοηθήσει στην διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας χωρίς να παρεμβαίνει στις αρμοδιότητες των κρατών μελών προτάσεις για μεγαλύτερη συνεργασία, για συνοριακή συνεργασία ε, όσον αφορά την ε, παροχή φαρμάκων, ε, τη συνταγογράφηση κλπ. με κινητά τηλέφωνα, το διαδίκτυο και την τηλεόραση μπορεί να επιτρέψει σε πολίτες ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση να έχουν πιο γρήγορη και καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Επίσης, ασθενείς με σπάνιες ασθένειες μπορούν να έχουν πρόσβαση σε ειδικά κέντρα σε όλη την Ευρώπη, γλιτώνοντας έτσι χρόνο, χρήμα και μετακινήσεις η έλλειψη διαλειτουργικότητας ανάμεσα στα ε, ηλεκτρονικά συστήματα που χρησιμοποιούν οι υπηρεσίες υγείας συχνά εντός της ίδιας χώρας, οι διαφορετικές χώρες, οι γλώσσες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, ε, μπορεί να αποτελέσουν προκλήσεις όσον αφορά την διασυνορική περίθαλψη. Οι προτάσεις για θέσπιση κοινών ε, ελάχιστων ε, προτύπων όσον αφορά τα δεδομένα μπορούν να οδηγήσουν σε καλύτερη λειτουργία και διαλειτουργικότητα των ε, ηλεκτρονικών υπηρεσιών υγείας, βελτιώνοντας την ασφάλεια των ασθενών. Επικροτούμε την έκκληση του εισηγητή και τώρα μερικές δικές μου παρατηρήσεις. Συμφωνώ απόλυτα με ε, την συνάδελφο ε, από τους σοσιαλιστές. Προέρχομαι από μια χώρα όπου προσπαθήσαμε να, έχουμε ψηφιακά στοιχεία για από την αρχή μέχρι το τέλος και είναι πάρα πολύ δύσκολο να λειτουργήσει ένα τέτοιο σύστημα. Και υπάρχει και κάτι ακόμα. Αν ε, κανείς είναι καλός hacker, δεν είναι δύσκολο να μπει κανείς να δει τι ασθένειες έχει ο κόσμος και να μπει στα προσωπικά του δεδομένα. Αυτό ήδη το έχουμε δει στη χώρα μου. Παρότι δεν είναι τόσο παλιές ε, αυτές οι παρότι δεν είναι τόσο παλιό αυτό το σύστημα των ψηφιακών πληροφοριών. Θα πρέπει λοιπόν να γνωρίζουμε πολύ καλά πώ θα το κάνουμε αυτό. Πιστεύω ότι υπάρχουν σημαντικέ δυνατότητε, ιδιαίτερα αν έχει κανεί σε μια σπάνια ασθένεια, ε, για την οποία υπάρχουν μόνο λίγοι καθηγητέ σε όλη την Ευρώπη που να μπορούν να ε, βοηθήσουν στην περίθαλψη. Αλλά πιστεύω ότι θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ την Άννα Ρόσπαχ. Δίνω το λόγο στην Κομισιόν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον αξιότιμο βουλευτή για την γνωμοδότηση του και ευχαριστώ και όλους τους βουλευτές που μίλησαν και στήριξαν την πρότασή μας, τουλάχιστον εγώ έτσι κατάλαβα. Ε, μερικά λόγια σχετικά με τα σχόλια που ακούστηκαν εκφράσατε κάποια αμφιβολία, κάποιο προβληματισμό για τις πράξεις κατεξοδότηση. Έχει υπάρξει ένα μνημόνιο κατανόηση ανάμεσα στο Κοινοβούλιο και την Κομισιόν. Αλλά σα εξηγήσω γιατί θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε ε, πράξη κατεξοδότηση. Όπω είπε η κυρία Μακάβαν, Αυτό αφορά το να είμαστε ικανοί σε 10 έτη να λάβουμε απόφαση για νέες προτεραιότητες. Είναι ένας τομέας αυτός ο οποίος κινείται πολύ γρήγορα. Ποτέ ε, είχαμε ακούσει το παρελθόν τις ε, ε, εταιρείε που υπάρχουν σήμερα, που έχουν ιδρυθεί και το ίδιο θα συμβεί τα επόμενα 5-10 χρόνια. Θα έχουμε λοιπόν ένα ευέλικτο μέσο, γι' αυτό χρειαζόμαστε λοιπόν τις ε, πράξεις κατεξοδότηση για να τροποποιούμε τα παρακτήματα. Έχουμε λοιπόν ανάγκη από ένα ευέλικτο εργαλείο. Τώρα σε ό,τι φορά το ζήτημα της μόχλευσης μπορώ εδώ να αναφέρω ερωτε... Ε, απαντήσεις προς την κυρία Αντωνέσκου και Μακάβαν αναφορικά με τα ε, περισσότερες πληροφορίες που θα πρέπει να χορηγηθούν για, τον, ε, <clears throat> τη μόχλευση. Θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε τα νέα χρηματοδοτικά μέσα, διότι θεωρούμε ότι σε περίπτωση, μάλλον σε καιρούς κρίσης και μείωση των κρατικών δαπανών, αυτός είναι ένας τρόπος για να προχωρήσουμε. Το ζήτημα της ε, κοινή ε, διευκόλυνση ε, τη χρηματοδότησή τη. Έχουμε προγράμματα 6 δι ε, ευρώ που θα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν. Μιλάμε γι' αυτό του είδου τη μόχλευση. Έχουμε, υπογρα... Έχουμε υπολογίσει περίπου 6 με 7 φορέ την τρέχουσα επένδυση και θα εξαπλαστεί, θα εξαπλαστεί δηλαδή θα επταπλιαστεί και θα μπουν περίπου 7 δις στο συνολικό πακέτο θα ανέρθει σε 50 εκατομμύρια ευρώ. Είναι πολλά, όπως ρώτησε ο αξιόμενος βουλευτής. Εμείς θεωρούμε ότι είναι πολύ λίγα. Αν θα μπορούσατε να διπλασιάσει τον προπολογισμό μας, θα ήμασταν ιδιαίτερα ευτυχείς. Έχουμε ένα χάσμα ε, περίπου 700 εκατομμυρίων. Λοιπόν, τα Θέλουμε να πετύχουμε τα 30 MB το 2020 και να φτάσει στο μεγαλύτερο δυνατό ποσοστό του πληθυσμού. Τώρα για το περιβάλλον έχουμε διάφορες υπηρεσίες που αναφέρονται στο παράρτημα και στοχεύουμε στο ζήτημα της, ε, ε, των εφιών μετρητών ένα παράδειγμα είναι αυτό. Και θα έχουμε σοβαρά αποτελέσματα στο τομέα της κατανάλωσης ε, ενέργειας αλλά και μείωσης της ρήπανσης. Νομίζω ότι κάλυψα τα περισσό, τις περισσότερες ερωτήσεις ε, που ετέθησαν. Ε, και αυτό θα κλείσω πώς ε, επιλέγουμε τα διάφορα προγράμματα που αυτό το παράδειγμα έχουμε τρεις διαφορετικούς τρόπους ε, για αυτό. Την διασυνοριακή σημασία, εάν έχει οριμάσει για ανάπτυξη και αν έχει ήδη, ε, έχουμε ήδη πειραματιστεί πάνω σε αυτό, αν έχει τύχει πιλωτικού προγράμματος. Ευχαριστώ. Φαίνεται λοιπόν πόσο αφορά αυτό το θέμα την Επιτροπή μας από πολλές πλευρές και για το περιβάλλον και για το κλίμα και για τα θέματα της υγεία. Αυτό με κάνει να πω ότι πρέπει να σκεφτούμε μήπως να καλέσουμε την Έλλη Κρούς εδώ στην Επιτροπή μας, την Επίτροπο που είναι αρμόδια για την ψηφιακή ατζέντα. Γιατί είναι πολλά τα θέματα που θα πρέπει και μπορούν να διεκπεραιωθούν από εκεί. γιατί είναι λίγο παιδί ε, αυτή η ιστορία και καλό θα ήταν να της δώσουμε μεγαλύτερη σημασία και όχι σε φτωχό συγγενή. Θα ήθελα να ξαναδώσω το λόγο στο συντάκτη νομοδότηση, στον κύριο Ρώση, παρακαλώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Εξαιρετική η πρότασή σας να καλέσουμε την κυρία Επίτροπο. Ευχαριστώ την Κομισιόν που ήταν σαφέστατη για κάποιες επιλογές όπως αυτή των ε, πράξεων κατεξοδότηση. Θα αξιολογήσουμε με τους ε, σκιώδεις τι θα πρέπει να κάνουμε. Εγώ όπως πάντα είμαι ανοιχτός στις τροπολογίες των συναδέλφων και θα αξιολογήσουμε το πώς ε, θα προχωρήσουμε περαιτέρω. Δύο απαντήσεις εντάχει να δώσω προς τη συνάδελφο Μακέβαν οποία είπε ότι τονίζουμε ιδιαίτερα την ε, θέμα της περίθαλψης και αυτή την απασχολεί το ζήτημα των ευαίσθητων δεδομένων. Ναι, είναι γεγονός. Εμείς ζητάμε να υπάρξουν ε, ε, παρόμοιοι κωδικοί ανάμεσα στα κράτη-μέλη για να αποφασίσουμε μέχρι πού μπορούμε να φτάσουμε για τα δεδομένα. Αυτό θα τα αποφασίσουν αυτοί που είναι και οι καταλληλότεροι. Ελπίζω να το κάνουμε εμείς. Τώρα, επειδή υπάρχει ελεύθερη διακίνηση, εκατομμύρια Ευρωπαίων πολιτών βρίσκονται σε διαφορετικούς χώρους και εδάφη σε σχέση με την επικράτεια της πατρίδας τους ε, και νομίζω ότι αν υπάρχει μια ε, ψηφιακή στήριξη που θα αναφέρει τις αλλεργίες, τις παθήσεις, την ε, ομάδα αίματος, ε, αν ανήκει ή όχι σε δωρητές οργάνων. Λοιπόν, αυτό ε, ε, σημαίνει πολλά. Μπορούμε με αυτόν τον τρόπο να σώσουμε ζωές. Δεν χρειάζεται ένα Ιταλό βρίσκεται στην Γαλλία ή ένα Γάλλο στην Αγγλία να μην υπάρχουν αυτέ τι πληροφορίε. Δεν νομίζω λοιπόν ότι οι hackers ε, θέλουν να γνωρίζουν αυτά τα στοιχεία. Τι του ενδιαφέρει η πάθηση ενό Ευρωπαίου πολίτη, τι του ενδιαφέρει αίματα αίματο. Δεν λοιπόν καίγονται για να μάθουν εάν κάποιο κινδυνεύει να πεθάνει αν του χορηγηθεί κάποιο φάρμακο αντί για κάποιο άλλο. Αυτό πρέπει να το ξέρει ο πολίτης και οι θεράποντες, οι ιατροί. Επίσης ασχοληθήκαμε με το θέμα ε, των σχέσεων με τη δημόσια δίκη. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό ζήτημα. Τώρα, τροπολογίες σχετικά με το περιβάλλον και επί ε, θεμάτων είναι ευπρόσδεκτες. Ευχαριστώ τη συνάδελφο Ρόσμπακ και αυτή έθιξε κάποιες, ε, κάποιους φόβους, κάποιες ανησυχίες, αλλά και εδώ είναι ζήτημα επιλογής τι θα μπούμε στα έγγραφα και στους ε, κώδικους Ε, υπενθυμίζω πως ε, υπάρχει ένα κείμενο που αφορά την διασυνορική περίθαλψη είναι γεγονός ότι οι πολλοί πολίτες πηγαίνουν για να για λόγους ε, ασθένειας, ε, αλλά μερικές φορές τη χάνει να ασθενήσουν όντας σε μια άλλη χώρα εκτός ε, της πατρίδας τους. Η συνάδελφος Αντωνέσκου αναφέρθηκε στην υποβολή τροπολογιών για το θέμα των προφοριών τα θέματα περιβάλλοντος και πρέπει να χρησιμοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους ε, διαθέσιμους πόρους και στη συνάδελφο Λίντα. Ευπρόσδεκτες ε, τροπολογίες για συγκεκριμένες προτεραιότητες σε σχέση με άλλους τομείς τώρα στη ε, συνεδρίαση των σκιωδών θα μπορούσαμε να το εμβαθύνουμε το θέμα. Αυτό που θα ήθελα να σας ζητήσω είναι να αποφασίζουμε τι θα κάνουμε σχετικά με τι ε, πράξει κατεξιοδότηση, να θέλουμε να διατηρήσουμε εμεί αρμοδιότητες ω κοινοβούλιο ή να τι αναθέσουμε στην Κομισιόν. Αλλά αυτό μπορούμε να το αποφασίσουμε ήχο και νυφαλίω όλοι μαζί. Ευχαριστώ προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών. Αύριο στις 12 το μεσημέρι θα ψηφίσουμε 25 και 26 Απριλίου. Στις 9 Μαρτίου είναι, συγγνώμη, η προθεσμία. Το Νοέμβριο θα ψηφίσει επί της ουσίας η Επιτροπή Βιομηχανίας από ό,τι βλέπω εδώ και στην Ολομέλεια το Γενάρη το 2013. Και um diese thematik, um diese thematik. Έχουμε χρόνο άπλετο στη διάθεσή μας, ε, ε, οπότε μπορούμε να το συζητήσουμε και με την αρμόδια επίτροπο, την κυρία Νέλη Κρούς, ενδεχομένω και άλλα θέματα. Έτσι, θα το σημειώσω στο ημερολόγιο μου στην ατζέντα μου. Ευχαριστώ. Πάμε στο επόμενο θέμα τώρα που είναι το σημείο 20. Εφαρμογή της οδηγίας πλαίσιο για τα απόβλητα. Συζήτηση, ανταλλαγή απόψεων με τους εκπροσώπους της Επιτροπής. Γκαρσία Μπούργκες. Πέρσι ε, πρότεινε να έρθει στην Επιτροπή μας να μας παρουσιάσει την εφαρμογή της οδηγίας, την πορεία της, την πρόοδο της και θα ακούσουμε τώρα ε, την ε, παρουσίαση του εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε και σας ευχαριστώ που μου δώσατε ε, χρόνο στην Επιτροπή σας για να σας κάνω αυτή την παρουσίαση για την οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα. Υποθέτω ότι γνωρίζετε ότι είναι ε, ακρογωνιαίος λίθος ε, της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και εφαρμογή της είναι πολύ δύσκολη ε, από τις πιο σοβαρές και δύσκολες ε, παραβιάσεις του κοινοτικού δικαίου είναι εκείνες που ε, αφορούν την οδηγία πλαίσιο για τα πόβλητα και υπάρχουν σοβαρά προβλήματα και λύματα στην εφαρμογή της. Αναφέρω ορισμένες βασικές απαιτήσει αυτής της οδηγίας. Θα σας πω για ποιες είναι οι προκλήσεις για την εφαρμογή ε, και δυσκολίες και στη συνέχεια θα σας παρουσιάσω τις δράσεις που προτιθέμεθα να αναλάβουμε. Um, ε, επιτρέψτε μου μερικά εισαγωγικά σχόλια. Πάρα πολύ σύντομα η εφαρμογή της νομοθεσίας περί αποβλήτων είναι κεντρικό ε, στοιχείο ε, της ατζέντα μας για την ε, αξιοποίηση των πόρων. Υπάρχει πολύ μεγάλος χώρος για δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Ο κύκλος συγγνώμη, ο κλάδος της ανακύκλωσης είναι πάρα πολύ ελπιδοφόρος και η πλήρη συμμόρφωση προς την κοινοτική νομοθεσία θα καταλήξει ε, σε δημιουργία 400.000 ε, νέων θέσεων απασχόλησης. Και επίσης θα μειωθούν σημαντικά οι εκπομπές ε, αερίων του θερμοκηπίου. Για να γίνουν όλα αυτά, θα πρέπει να υπάρχει πλήρης συμμόρφωση με την κοινοτική νομοθεσία. Αυτό θα σήμαινε ότι μπορούμε να αποφύγουμε εκπομπές ε, ρήπου αντίστοιχους με εκείνους που εκπέμπουν 47 εκατομμύρια αυτοκίνητα. Είναι γενική οδηγία αυτή που ε, ρυθμίζει θέματα ε, που δεν εμπίπτουν σε ειδική νομοθεσία όπως αφορά τα ε, παλαιά οχήματα ή ε, τα ηλεκτρονικά συσκευές. Εγώ θα αναφερθώ μόνο στα αστικά απόβλητα. Γιατί, γιατί από ποσότητας, από πλευράς ποσότητας είναι από το μεγαλύτερο όγκο, το 1 τρίτο είναι των αστικών αποβλήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, είναι ένας κάλλιστος τρόπος να μετρήσουμε τις επιδόσεις των κρατών μελών. Τα δημοτικά απόβληματα, απόβλητα Ε, και είναι πιο εύκολο να αξιολογήσουμε και να μετρήσουμε τις στατιστικές σε σχέση με τα ε, απόβλητα της γεωργίας ή της βιομηχανίας. Είναι πάρα πολύ περίπλοκη η νομοθεσία και αρκετά ευρεία. Ε, θα αναφερθώ σε δύο βασικές διατάξεις. Η ιεράρχηση των αποβλήτων και στόχος πρόληψης. θα πρέπει να γίνουν επιλογές για τη διαχείριση των αποβλήτων στα κράτη-μέλη. Η πρόληψη βεβαίω είναι η καλύτερη επιλογή. Ε, μετά είναι η ανακύκλωση, η επανάκτηση και τελικά είναι η διάθεση ε, στους ε, η αποτέφρωση, ε, η κάψη των σκουπιδιών. Αυτή είναι η καψη των σκουπιδιων αυτο επιλογή και η έσχατη και η χειρότερη προφανώς. Έχουμε στόχο ανακύκλωσης που αφορά ιδίως τα νοικοκυριά και τα δημοτικά απόβλητα. Είναι πάρα πολύ ε, δεσμευτικός αυτός ο στόχος. Ε, είναι περίπλοκη όμως η νομοθεσία στην οδηγία και η διατύπωση. Αφορά τα κράτη-μέλη και τα ε, υποχρεώνει να ανακυκλώνουν το 40% των αποβλήτων Ε, είχα προετοιμάσει διαφάνειες με τις στατιστικές για την κατάσταση το 2009. Αλλά δυστυχώς υπάρχουν τεχνικά προβλήματα. θα σα δώσω σε όλους του βουλευτέ τη παρόντης στην αντίγραφα, γιατί δεν λειτουργεί το μηχάνημα για τα slides. Οι ε, διαφάνειες λοιπόν αυτές δείχνουν ε, τα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι υπηρεσίες της Eurostat και η κατάσταση είναι άκρο ανησυχητική. Το 2009 οι χωματερές, και επαναλαμβάνω χωματερές, τα που είναι η χειρότερη επιλογή, ε, στην ιεράρχηση της, της διαχείρισης των αποβλήτων μάλλον, παραμένει το βασικό σύστημα διαχείρισης των αποβλήτων στην Ένωση. 38% του συνόλου των δημοτικών αποβλήτων ε, θάβονται σε χωματορές και... Σε ό,τι αφορά ε, την ανακύκλωση ήταν πολύ μακριά από το στόχο του 50%. 42% όλων των αστικών αποβλήτων των ανακυκλωνόταν το 2009. Αυτό που μας ανησυχεί περισσότερο είναι ότι οι στατιστικές δείχνουν μεγάλες αποκλίσεις στις επιδόσεις των κρατών μελών. Μπορούμε να κάνουμε διακρισία ανάμεσα σε τρεις ομάδες κρατών μελών. Πρώτα απ' όλα έχουμε μία ομάδα των καλών μαθητών που είναι κάτω από 20% η διάθεση σε χιτά και να κτίσει πάνω από 80%. Βέλγιο, Δανία, Γερμανία, Λουξεμβούργο, κάτω χώρες, ε, Αυστρία, Σουηδία είναι η ομάδα των κρατών αυτών. Και ε, βασικά οι χώρες αυτές δεν θα πρέπει να έχουν μεγάλα προβλήματα στην ιεράρχηση των αποβλήτων και ε, στο να καταφέρουν να φτάσουν στους στόχους της ανακύκλωσης. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι ορισμένα κράτη-μέλη σε αυτή την ομάδα έχουν αναπτύξει υπεραποτέφρωση και αυτό μπορεί να είναι εις βάρος της ανακύκλωσης. Ε, στη συνέχεια ακολουθεί μια ομάδα με τρίων επιδόσεων με χίτα 20 με 65% Ισπανία, Γαλλία, Ιρλανδία, Ιταλία, Φινλανδία, Πορτογαλία, Σλοβενία και Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτές οι χώρες σίγουρα θα πρέπει να κάνουν πια προσπάθεια να αναβαθμίσουν τα συστήματα ανακύκλωσης και διαχείρισης των αποβλήτων και ιεράρχησης. Επιπλέον ε, θα πρέπει να ξεπεράσουν κάποια τοπικά και περιφερειακά προβλήματα μεγάλη σημασία και πολύ ε, οξέα πολλές φορές. Και τέλος, έχουμε μια ομάδα κρατών που είναι κακές οι χώρες επιδόσεις και δεν θα σας εκπλήξει ότι εκεί θα βρούμε όλες τις νέες χώρες, τις 12, με εξαίρεση τη Σλοβενία, συν ένα άλλο κράτος μέλος που δείχνει επίπεδα επιδόσεων τόσο κακά ε, όσο είναι οι Σαχθέντες Και η χώρα αυτή είναι η Ελλάδα. Πάνω από 75% είναι ηχητά και καταρχήν οι χώρες αυτές θα χρειαστούν δραματικό επανασχεδιασμό του τρόπου διαχείρισης των αποβλήτων και των συστημάτων για να ξεφύγουν από την υπερβολική εξάρτηση ε, από την διάθεση χιτά και να περάσουν σε ανακύκλωση γιατί είναι πολύ χαμηλή. Τώρα, τι ε, θα πρέπει να κάνουμε για να κλείσει αυτό το χάσμα εφαρμογή. Προφανώ, μαγική λύση δεν υπάρχει και πανάκια. Ε, ε, υπάρχουν όμως πολλές δράσεις, κλειδιά που ήδη έχουν αναλυφθεί. Η οδηγία θα πρέπει να μεταφερθεί και να εφαρμοστεί σωστά σε όλα τα κράτη-μέλη. Αυτό είναι το βασικό και το κυριότερο. Το Δεκέμβρη του 10 έχει λήξει η προθεσμία, αλλά δυστυχώς ε, ε, πολλά κράτη-μέλη ακόμα δεν έχουν μεταφέρει στο εθνικό του δίκαιο ε, την οδηγία. Έχουμε προσφύγει επί παραβάση και ελπίζουμε όλα τα κράτη-μέλη να συμμορφωθούν σύντομα. Στη συνέχεια θα πρέπει να ελέγξουμε τι γίνεται με τα μέτρα μεταφοράς και υλοποίησης αν συμμορφώνονται πλήρως με την οδηγία. Αυτό θα το κάνουμε το δεύτερο εξάμεινο του 12 και αν χρειαστεί θα ξεκινήσουμε διαδικασίες επί παραβιάση το 2013. Εκτός από τη μεταφορά της οδηγίας, τα κράτη-μέλη οφείλουν να εγκρίνουν σχέδια διαχείρισης αποβλήτων και προγράμματα πρόληψης παραγωγής αποβλήτων, έτσι ώστε να εφαρμόσουν σωστά την οδηγία. Γι' αυτό θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ελέγξει τα προγράμματα ε, και τα σχέδια. Δυστυχώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει αυτή τη δυνατότητα ε, στις υπηρεσίες της. Για τα προγράμματα αυτά, διότι πολύ συχνά ε, εγκρίνονται σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, όχι σε εθνικό και θα πρέπει να ελέγχουμε εκατοντάδες προγραμμάτων. Γι' αυτό αναλύουμε διάφορες δυνατότητες για να μπορέσουμε καλύτερα να ελέγξουμε. Ε, δημιουργία ενός ευρωπαϊκού οργανισμού αποβλήτων ήταν μία από τις επιλογές αυτές, αλλά καταλήξαμε ότι θα ήταν πιο απλό αλλά και πιο αποτελεσματικό να επαφιέμεθα σε ένα οργανισμό που ήδη υπάρχει, που είναι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος συνεργαζόμαστε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μαζί του για να ε, αναπτύξουμε ένα μοντέλο που θα μας βοηθήσει να αξιολογήσουμε τις προτάσεις και τα σχέδια των κρατών μελών. Επίσης, ε, εκπονούμε οδηγίες καθοδήγησης, κατευθυντήριες γραμμές για τη διάδοση ε, και των βέλτιστων πρακτικών. Όλα τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας δείχνουν ότι το σύστημα το ρηπαίνων πληρώνει ε, και, ε, δηλαδή με μια επιβολή τελών όσο περισσότερα ε, απόβλητα παράγει κανείς τόσο περισσότερα πληρώνει, είναι αποτελεσματικά. Η εμπειρία στα κράτη-μέλη με τις καλύτερες επιδόσεις είναι πολύ σαφής προς την κατεύθυνση αυτή. Τώρα ολοκληρώνουμε μια μελέτη για αυτό το θέμα και θα προσπαθήσουμε να οθήσουμε τα κράτη-μέλη που είναι σε χαμηλότερες επιδόσεις να χρησιμοποιήσουν τα οικονομικά μέσα πιο εντατικά και είναι επίσης ενδιαφέρον να καταλάβουμε ότι σε ε, περίοδους οικονομικής κρίσης και δημοσιονομικής λιτότητας η χρήση οικονομικών μέσων για την διάθεση των αποβλήτων μπορεί να αποτελέσει επιπλέον πηγή εισοδήματο για τους Δήμους και τις κοινότητες. Τέλος, είναι σαφές ότι η κοινοτική χρηματοδότηση και ιδιαίτερα αυτό το Ταμείο Συνοχής και το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης μπορεί ε, να παίξουν ένα ρόλο κλειδί στην αναβάθμιση των συστημάτων διαχείριση αποβλήτων στις χώρες με τις χαμηλότερες επιδόσεις. Γι' αυτό θα πρέπει οπωσδήποτε να βεβαιωθούμε ότι οι πορεί χρησιμοποιούνται για αυτό το συγκεκριμένο σκοπό για να βελτιωθεί η διαχείριση των αποβλήτων και επίσης είναι σημαντικό να πιάνουν τόπο τα χρήματα και να ε, εφαρμόζεται καλύτερα κοινοτική νομοθεσία περί αποβλήτων. Όπως ε, ε, λέει και ο δικός χάρτης, θα πρέπει να αφιερώνεται τα κονδύλια σε προγράμματα υψηλής ποιότητας και όχι στη δημιουργία νέων χιτά. Για τις επόμενες χρονιές, την επόμενη περίοδο των δημοσιονομικών προοπτικών θα πρέπει να ελέγχουμε εκ των προτέρων τα σχέδια που υποβάλλονται εάν εντάσσονται στο σύστημα ε, διαχείρισης αποβλήτων που συνάδει με την κοινοτική νομοθεσία. Τελειώνω εδώ με αυτό την παρουσίασή μου. Έχω φτάσει στο τέλος. Δεν ξέρω θέλετε να συνεχίσω τώρα να απαντήσω στις ερωτήσεις που έχουν ήδη υποβληθεί γραπτός. Με χαρά να το κάνω. Θέλετε να συνεχίσω? Μάλιστα. Ε, προς το παρόν μια στιγμή. Ευχαριστώ πολύ για την εκτενή σας παρουσίαση και την εξαντλητική. Έχουμε και προφορικές ενδιάμεσες ερωτήσεις, θα τις πάμε για να έχετε την ευκαιρία να τις απαντήσετε. Η Άννα Ρόσμπαχ και μετά Φλόρεντς και μετά Χάουγκ και πάει λέγοντας. Ο Ρίχαρτ Ζέμπερ, Ευχαριστώ πολύ για ε, την σαφή παρουσίασή σας και μας δώσατε μια, μια σαφή εικόνα, μια ακριβή εικόνα για το εγγύς μέλλον. Αυτό είναι σημαντικό. Εγώ προέρχομαι από τη Δανία. Είμαστε λοιπόν ένα από τα καλά παιδιά της τάξης, από τους καλούς μαθητές. Ε, Πιστεύω λοιπόν ότι τα απόβλητα δεν είναι απόβλητα, είναι ένας ε, σημαντικός πόρος. Έχω λοιπόν μια ερώτηση προς εσάς. Τι πιστεύει η Κομισιόν όσον αφορά την αποτελεσματικότητα ή η έλλειψη αυτής σε κάποιες χώρες ε, την αποτελεσματικότητα της οδηγίας, για τα, της οδηγίας για τα απόβλητα για τα θαλάσσια απόβλητα και πώς μπορούμε να σταματήσουμε τη μεταφορά αυτών μέσω των ποταμών ε, στους ωκεανούς. Η Κομισιόν πώς βλέπει την ε, περαιτέρω εφαρμογή της οδηγίας σε σχέση με ε, την εστίαση σε περισσότερη ανακύκλωση και πώς βλέπει τα απόβλητα ως πόρο ιδιαίτερα στις, ε, στα νέα κράτη. Ευχαριστώ Άννα Ρόσπαχ, ο Καρλ Χάινς Φλόρενς και κατόπιν η Γιούτα Χάουκ. Ε, ήθελα να ε, σας παραπέμψω στην γραπτή μου ερώτηση. Παρακαλώ να μου απαντήσετε. Ε, ευχαριστώ, Ιούτα Χάουκ. Ήθελα να αναφερθώ στην ε, δήλωση του ε, προσώπου της Κομισιόν που είπε ότι θα ήταν χρήσιμο να έχουμε μια υπηρεσία για τα απόβλητα. Η Κομισιόν έχει ήδη νομική, ετοιμάζει νομική βάση για αυτόν τον οργανισμό, ε, διότι χρειαζόμαστε μια σωστή πρόταση. Ή ή προβλέπει ε, τροποποίηση ε, της εντολής για, για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος. Και ε, πιστεύω ότι η Κομισιόν όσον αφορά το ρόλο της που είναι να κάνει τον αστυνομικό ε, όσον αφορά την εφαρμογή της νομοθεσίας ε, περί αποβλήτων στην, ε, στα κράτη-μέλη την κοπανάει, δεν πληρεί τα καθήκοντά της και θέλει να, να δημιουργήσει έναν οργανισμό που θα κάνει τη δουλειά αντί για αυτήν. Ευχαριστώ πολύ Γιούτα Χάουκ. Ο Ρίχαρτ Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Μπορώ να συμφωνήσω με την Γιούτα το να δημιουργήσουμε πάλι ειδικό οργανισμό, δεν ξέρω. Θα ήθελα να ρωτήσω την Κομισιόν ε, τι έχει κάνει μέχρι τώρα για να στηρίξει τα κράτη-μέλη κατά την εκπλήρωση των στόχων αυτών που έχουν τεθεί από κοινού. Από πρακτικής πλευράς και από τεχνικής πλευράς. Μήπως θα έπρεπε να δημιουργήσουμε δίκτυα ώστε να μάθει ο ένας από τον άλλον, όπως συμβαίνει και σε άλλους τομείς που συνδέονται με το περιβάλλον. η έκκληση της Κομισιόν να δοθούν ε, χρήματα από τα περιφερειακά ταμεία ε, και τα εθνικά ταμεία είναι ε, σωστή, αλλά όσον αφορά τα χειρότερα κράτη εδώ, την Βουλγαρία και την Ρουμανία, στις χώρες αυτές δεν υπάρχει εξάρτηση των πόρων, δεν υπάρχει απορρόφηση των πόρων. Θα ήθελα λοιπόν η Κομισιόν να μου πει μήπως θα μπορούσαν να συνεργαστούν με τις ε, συναδέλφους τους από την Γενική Διεύθυνση Ρέγγι ε, και να εξετάσει αυτό το θέμα της ε, συγχρηματοδότησης στις χώρες. Και η Ελλάδα παίρνει χρήματα, αλλά πρέπει να ε, συγχρηματοδοτήσει, το οποίο σημαίνει ότι ε, μεγάλα ποσά δεν εξαντλούνται και ε, απαιτεί ο κόσμος οργανισμό. Εγώ δεν καταλαβαίνω τι θα πρέπει να κάνει ο οργανισμός αυτός. Θα πρέπει να δούμε τι μπορούν να πετύχουν οι δύο επίτροποι, ο Χάν και ο Πτότσνικ, στο θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, Ρίχαρτ. Τον λόγο έχει ο κύριο Χρυσόγελο και μετά η κυρία Μάρκου Νάιτ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα μιλήσω και εκ μέρους της ομάδας των Πράσινων στα επόμενα θέματα. Ε, ήθελα να ε, πω ότι προέρχομαι από μια χώρα που είναι από τους κακούς μαθητές δυστυχώς στο θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων και προσωπικά έχω ασχοληθεί πάρα πολύ. Ε, ήθελα να πω ε, κατά πόσο η Κομισιόν ε, βλέπει ότι σε μια περίοδο που είναι μεγάλη οικονομική κρίση μπορούν να χρηματοδοτούνται ακόμα σχέδια τα οποία δεν εφαρμόζουν αφενός την ιεράρχηση που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Οδηγία, την ιεράρχηση στις μεθόδους διαχείρισης των απορριμμάτων που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Οδηγία και απ' την άλλη επιλέγονται οι πιο δαπανηρές μέθοδοι όπως στην περίπτωση της Αττικής αν έχει να σχολιάσει κάτι τέτοιο. Και το δεύτερο είναι ότι στο παρελθόν έχουν χρηματοδοτηθεί πάρα πολλά έργα κατασκευή χιτά, ενώ θα έπρεπε να υπάρχει δέσμευση με βάση και τη συμφωνία που είχε γίνει από το 2002 ήδη ε, τα έργα που προωθούνται με χρηματοδότηση ευρωπαϊκή να ακολουθούν την ιεραρχία, δηλαδή την πρόληψη, ε, επαναξενοποίηση, ανακύκλωση κλπ. Έχουμε δει πολλές φορές να γίνονται χώροι υγειονομική ταφή χιτά χωρίς να προηγούνται όλες οι άλλες μέθοδοι και αν ε, σκοπεύει να κάνει κάτι η Κομισιόν σε σχέση με το θέμα αυτό. Να ευχαριστήσω την Κομισιόν για την παρουσίαση. Εγώ είμαι Λιθουανή. Είμαι λοιπόν από μια χώρα που δεν τα πάει και τόσο καλά σε ορυφά διαχείριση των ε, αποβλήτων. Λυπάμαι που βλέπω αυτά τα στοιχεία, αλλά πάρα πολλές συζητήσεις διεξάγονται στην χώρα μου σκεφτόμαστε για ποιο λόγο το σύστημα δεν λειτουργεί αποτελεσματικά. Και θα ήθελα να ρωτήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι ερωτήσεις λαμβάνεται από αυτές τις 12 χώρες μέλη για την διαχείριση. Υπάρχουν ενδεχόμενα συστημικά προβλήματα. Ποια είναι τα επιχειρήματα λοιπόν τα οποία καταθέτουν τα κράτη-μέλη, για ποιο λόγο δεν καταφέρουν να ε, ε, υλοποιήσουν το σύστημα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δύο ερωτήσεις θα είχα εγώ προς τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ερώτηση πρώτη. Τι γίνεται με το λαθρεμπόριο και τις λαθρές εξαγωγές ε, απορριμμάτων. Κάνατε ήδη μια έρευνα σε 22 κράτη-μέλη και ορισμένα γειτονικά κράτη επίσης. Επιπλέον, γράψατε σε μια άλλη έκθεση ότι υπάρχει διασύνοριακό εμπόριο αποβλήτων και μάλιστα λαθρεμπόριο. Ε, η μία στις πέντε μεταφορές είναι λαθρέα, το 20%. Τι έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα προηγούμενα χρόνια και τι προτίστε να κάνει τα επόμενα. Έχετε εκπονήσει καμία πρόταση. Γιατί αυτή η έκθεση δημοσιεύτηκε πέρυσι. Και επίσης γράφει ότι από ό,τι φαίνεται στα περισσότερα κράτη-μέλη το επίπεδο παραγωγής απορριμμάτων είτε είναι σταθερό είτε αυξάνει. Στα 27 κράτη-μέλη από το 2006 έως το 2008 είχαν μειώσει την παραγωγή αποβλήτων κατά 10% αλλά στη συνέχεια αυξήθηκε. Αυτές οι μεταβολές που οφείλονται, είναι τυχές, είναι καλύτερη πρόληψη, οφείλεται η οικονομική κρίση. Αυτές τις ερωτήσεις που κάνατε και γράφετε στις εκθέσεις σας τις έχετε απαντήσει. Έχετε κανένα σχέδιο για το μέλλον, για την πρόληψη παραγωγής απορριμμάτων και λιμάτων. Και τι προτείνετε για το μέλλον. Ευχαριστώ. Η Φρίντα Μπρέπουλς. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Χαίρομαι που έχουμε και πάλι τα στοιχεία, τα αριθμητικά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αν θυμάμαι καλά, πριν από μερικά χρόνια για την αναθεώρηση της οδηγίας αποβλήτων είχαμε συζητήσει και τα είχαμε ξαναπεί αυτά. Και είχαμε δει τα 10 νέα κράτη-μέλη ε, που ζητούσαν ε, προθεσμία για να φτάσουν σε κάποιους στόχους και την έλαβαν. 7 χώρες, παλιές εντός εισαγωγικών, είναι κάτω του μέσου όρου. Τώρα βλέπω για Ελλάδα, Ισπανία, Πορτογαλία, Ιταλία και Ιρλανδία. Ακριβώς χώρες που έχουν κακές επιδόσεις. Είπατε εισαγωγικά ότι κανονικά θα πρέπει να έχουν εφαρμόσει πλήρως την οδηγία και να την έχουν μεταφέρει. Και μάλιστα αυτό θα δημιουργούσε πάνω από 400.000 νέες θέσεις εργασίας και διερωτώ με, καλά τι περιμένουν αυτέ οι χώρε, ποιο είναι το πρόβλημα. Ορίστε, χρειάζονται και νέε θέσει εργασία, ακριβώ οι ίδιες χώρες, αλλά αδρανούν, δεν εφαρμόζουν την οδηγία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μα λέει, ωραία, θα βγάλουμε κάτι εφητήριε γραμμέ, βέλτιστες πρακτικέ, διάδοση. Ήδη από το 70 στη Φλάδρα έχουμε καταλήψει τις χωματερές και τους χιτά. Μα πώς είναι δυνατόν οι άλλες χώρες δεν το καταλαβαίνουν, δεν μπορούν να υποχρεωθούν με τον ΑΒ τρόπο να λάβουν αυτά τα μέτρα. Και ρωτώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχετε περιφερειακές στατιστικές για το Βέλγιο ας πούμε, έχουμε χωριστά στη Φλάντρα και στη ε, Βαλονία αρμοδιότητες είναι αρμοδιότητα της περιφέρειας ε, το περιβάλλον και αυτά τα θέματα και η νομοθεσία. Έχετε αυτά τα περιφερειακά στοιχεία για το Βέλγιο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Μπρέπουλς. Ο κύριος Γκερμπράντι, τελευταίος. Ευχαριστώ πρόεδρε. Έχω μια ερώτηση που έχει να κάνει με το ρόλο του ιδιωτικού τομέα στη διαχείριση των αποβλήτων με την αύξηση των τιμών των πόρων βλέπουμε ότι τα απόβλητα θεωρούνται όλο και περισσότερο πολύτιμος πόρος αντί για κάτι το οποίο πρέπει να ξεφορτωθούμε. Υπάρχουν τεράστιες επενδύσεις. Οι επενδυτές ε, εστιάζουν στην ε, βιομηχανία ανακύκλωσης. Υπάρχουν λοιπόν σημαντικές ευκαιρίες και φαντάζομαι ότι κάτι τέτοιο θα επιταχύνει την διαδικασία εφαρμογής της νομοθεσίας Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα απόβλητα και αναρωτιέμαι τι κάνει η Κομισιόν για να κινητοποιήσει τον ιδιωτικό τομέα και αν η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων επίσης συμμετέχει, διότι συχνά απαιτούνται σημαντικές επενδύσεις για να δημιουργηθούν οι χιλιάδες θέσεων απασχόλησης που ε, περιμένουν να δημιουργηθούν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ να δώσω τον λόγο στην Κομισιόν για να απαντήσει. Uh, Ευχαριστώ, θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Έχω εδώ ένα μακρύ κατάλογο από ερωτήσεις. Θα προσπαθήσω να τις απαντήσω με τη σειρά με την οποία ετέθησαν και ελπίζω πως δεν θα κάνω λάθη. Τα πρώτη ερώτηση από την κυρία Ρόσμπαχ για τη θαλάσσια ρήπανση. Αυτό συνδέεται με την κακή εφαρμογή της νομοθεσίας περί απορριμμάτων. Φυσικά και ναι, το πρόβλημα είναι ότι υπάρχουν απορρίμματα που για τον ένα ή τον άλλο λόγο διαφεύγουν άπορα τα συστήματα διαχείρισης και καταλήγουν στο θαλάσσιο περιβάλλον μέσω καλύτερης εφαρμογής ε, της νομοθεσίας ε, περί απορρίπτων μπορούμε να συμβάλλουμε στην επίλυση του προβλήματος ε, της θαλάσσιας ρήπανσης. Μία άλλη ερώτηση σχετικά με το δυναμικό, δυναμικότητα μάλλον του συστήματος διαχείρισης των απορριμμάτων ήδη είπα στην παρουσίασή μου πως ε, η εφαρμογή της νομοθεσίας ε, περί απορριμμάτων είναι ουσιώδες ε, στοιχείο της ατζέντα μας για την διαχείριση των πόρων. Εκτιμούμε ότι οι εξοικονομήσεις θα ανέλθουν σε 72 εκατομμύρια ευρώ ετησίως σημαντικό ποσό. Ο κύριος Φλόρενς αναφέρθηκε στις ερωτήσεις που έχει καταθέσει. Η πρώτη αφορά την ιεράρχηση των αποβλήτων και το πώς εφαρμόζεται από τα κράτη-μέλη από τη στιγμή της μεταφοράς του στην Εθνική Νομοθεσία. Υπάρχουν όντως ε, κάποια προβλήματα. Ήρθαμε σε επαφή με ορισμένα κράτη-μέλη και όπως είπα και στην παρουσίασή μου κάνουμε έναν έλεγχο πλήρους συμμόρφωσης ε, σχετικά με τη ε, μέτρα μεταφοράς, ε, κάτι το οποίο θα ξεκινήσει αργότερα μέσα στο έτος. Και ενδεχόμενα να προβούμε σε προσφυγή επί παραβάση. Τώρα, η δεύτερη όρεντς αφορά στην αυτάρκεια και τον ε, ανταγωνισμό ανάμεσα στα νομικά πρόσωπα υποδημόσιο έλεγχο και τον ε, ιδιωτικό κλάδο. Δεν προβλέπονται συγκεκριμένε διατάξεις ε, επί του θέματος, αλλά οι συνάδελφοι στην Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού ερευνούν εάν κανόνες ε, που υπάρχουν στα κράτη-μέλη συμμορφώνονται με την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ζητήματα ανταγωνισμού. Η επόμενη ερώτηση αφορά την υπηρεσία απορριμμάτων. Στην παρουσίασή μου είπα ότι αυτή τη στιγμή μέχρι τώρα δεν ε, έχει προβλεφθεί η σύσταση ενός ε, νέου σώματος, νέου φορέα. Πρόθεσή μας ε, είναι να συνεργαστούμε με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Περιβάλλοντος. Την αυτή ερώτηση έρχεται η κυρία Χάουγκ. Δεν προτιθέμεθα, δεν προβλέπουμε ούτε μία αλλαγή στον κανονισμό που προβλέπει τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος πιστεύουμε ότι σύμφωνα με την εντολή της η υπηρεσία μπορεί να ε, να παρακολουθεί τις ε, εξελίξεις της στα κράτη-μέλη και αυτή η δουλειά της θα μας βοηθήσει κατά την άσκηση των καθηκόντων μας, ε, ενεργώντας ως θεματοφύλακες των συνδικών αναφορικά με, με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και δεν προτιθέμεθα να αναθέσουμε αυτή την, αυτό το έργο σε κάποιον άλλο οργανισμό, σε κάποιον άλλο φορέα. Και μια άλλη ερώτηση σχετικά με το ότι πράττει η Κομισιόν προκειμένου να διασφαλίσει ότι περισσότερο οι πόροι χρησιμοποιούνται για την στήριξη της διαχείρισης ε, απορριμμάτων στα κράτη-μέλη. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω πως ε, εργαζόμαστε στενά με την Γενική Διεύθυνση Ρίτζο προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι περισσότερα κονδύλια χρησιμοποιούνται για την εφαρμογή της ε, οδηγίας ε, περί απορριμμάτων και πιστεύω ότι θα πετύχουμε κάποια πρόοδο στο ζήτημα ερώτηση του κυρίου Χρυσόγελου σχετικά με την κατάσταση στην Ελλάδα. Η Ελλάδα περιλαμβάνεται μεταξύ των ε, χειροτέρων μαθητών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κρίνουμε πως ε, θα πρέπει να επανεξετάσουμε το ζήτημα των χιτά και δεν θεωρούμε μακροπρόθεσμα ότι άλλες επιλογές πέραν της ε, των χιτά θα είναι πιο δαπανηρές. Αυτό που θα πρέπει να γίνει είναι να μην σπαταλάμε πόρους Μία άλλη ερώτηση από την κυρία Μορκουνάιτε γιατί τα νέα κράτη-μέλη αντιμετωπίζουν δυσκολίες ε, κατά την εφαρμογή της ε, νομοθεσίας ε, περί απορριμμάτων για τα νέα, νέα κράτη-μέλη αυτό αποτελεί νέα πρόκληση. Τα κράτη-μέλη τα οποία τώρα είναι τα πιο αποτελεσματικά να ξέρετε ότι Χρειάστηκαν 20 έτη για να φτάσουν στη σημερινή κατάσταση. Τα νέα κρατημέλη δεν ε, έχουν 20 έτη, απλά θα πρέπει να υποφεληθούν από την εμπειρία των άλλων κρατών μελών και κρίνω ότι με την στήριξη και την οικονομική βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα καταστεί δυνατόν να προχωρήσουν αρκετά γρήγορα. Η Eurostat ε, ήδη ε, παράγει κάποιες στατιστικές ενημερωμένες, επικαιροποιημένες για τη διαχείριση των ε, απορριμμάτων και φαίνεται ότι μέσα σε ένα χρόνο κάποια νέα κράτη-μέλη όπως Πολωνία, Σλοβακία πέτυχαν σημαντική πρόοδο αυξάνοντας ε, το ποσοστό ανακύκλωσης. There was a question by Μια άλλη ερώτηση τώρα. But to be very frank, ε, I ε, cannot read my notes. Αλλά εδώ πραγματικά δεν μπορώ να διαβάσω τις σημειώσεις μου. Θα περάσω στην επόμενη ερώτηση και αν ο κύριος Άβερ επιθυμεί μπορεί να μου ξαναθέσει το ερώτημα. Ε, η κυρία Μπρέπολς. γιατί η κατάσταση είναι, συνεχίζει να είναι κακή σε κάποια κράτη-μέλη. Ναι, υπάρχουν παλιά κράτη-μέλη ε, χώρες ε, που δεν τα πάνε και τόσο καλά, αλλά θα πρέπει να ξέρετε ότι η οδηγία αυτή είναι καινούρια, η προθεσμία για μεταφορά της οδηγίας ε, σε εθνική νομοθεσία εξέπνευσε το 2010 και δεν υπήρχαν κάποιοι συγκεκριμένοι στόχοι, δεν υπήρχε ε, κάποια δεσμευτική ιεράρχηση. Επίσης έθεσε και μια άλλη ερώτηση για τις περιφερειακές στατιστικές για ορισμένα κράτη-μέλη και δι για το Βέλγιο. Ξέρουμε ότι η Φλάνδρα και η Βαλονία ε, αναφέρουν χωριστά, αλλά άλλα κράτη-μέλη, ακόμα και αν έχουν περιφερειακή δομή, οι ε, στατιστικές υποβάλλονται ε, τρόπο, με τρόπο παγιωμένο. Και τέλος, ε, τι πράττουμε για να παροτρύνουμε τον ιδιωτικό τομέα. Έχουμε την εντύπωση πως ο ιδιωτικός τομέας δεν χρειάζεται να τύχει ιδιαίτερη παρότρεση ιδιαίτερων κινήτρων, διότι η διαχείριση των αποβλήτων και των απορριμμάτων ε, είναι business. Εμείς θέλουμε να έχουμε ένα καλό ρυθμιστικό περιβάλλον, ένα, μια κατάλληλη πολιτική και πιστεύουμε ότι το καλύτερο πράγμα που μπορούμε να προσφέρουμε για να στηρίξουμε τον ιδιωτικό τομέα είναι να διασφαλίσουμε πως ε, η οδηγία πλαίσιο εφαρμόζεται ορθά. Ευχαριστώ πολύ. Θα ξαναδώσω το λόγο στον κύριο Αντζαχιόνερ για να κάνει την ερώτησή του ξανά. Ε, ε, Ευχαριστώ. Είναι Τώρα για μένα, σαν διαγώνισμα ως πολιτικό, να ξανακάνω, μου ζητάτε την ίδια ερώτηση δύο φορές. Δύο ερωτήσεις έκανα και τώρα θα πρέπει να τις ξαναθυμηθώ ακριβώς τις ίδιες. η πρώτη ερώτηση ήταν, ποια μέτρα προτίθεται να λάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να αντιμετωπίσει το θέμα ε, του λαθρεμπορίου, του διασυνοριακού αποβλήτων και αν έχετε κάνει αναλύσεις στα 22 κράτη-μέλη που κάνατε την έρευνα, σε τι συμπέρασμα οδηγηθήκατε. Βρήκατε ότι το 20% ε, των μεταφορών αποβλήτων ε, είναι παράνομες των διασυνοριακών. Το ξέρετε αυτό και τι θα κάνετε για να το αντιμετωπίσετε. Πέρσι το Γενάρη δημοσιεύσατε αυτή την έκθεση για την ε, παραγωγή αποβλήτων και την επανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση και διαπιστώσατε ότι στα περισσότερα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυξάνεται η παραγωγή αποβλήτων. Συνεχώς. ενώ από το 2006 έως το 2008 είχε μειωθεί κατά 10% ε, λόγω της ε, καλής επίδοσης κάποιων ε, συγκεκριμένων κρατών. Δεν σημαίνει ότι μειώθηκε παντού το ίδιο. Σε άλλες χώρες αυξάνεται η παραγωγή αποβλήτων και είπατε ότι χρειάζεται και περαιτέρω ανάλυση κτλ. Την έχετε κάνει την ανάλυση αυτή γιατί μειώθηκε η παραγωγή αποβλήτων σε ορισμένες χώρες, επειδή συμμορφώθηκαν, επειδή περιορίστηκε η κατανάλωση λόγω της οικονομικής κρίσης λόγω πρόληψης. Είναι μια ερώτηση που γράψατε στην περσινή σας έκθεση και προβληματίζεστε, κάνετε ερωτήσεις η ίδια Επιτροπή προς τον εαυτό της. Τις έχετε απαντήσει αυτές. Ε, η Γιούτα παρακαλώ. Ζητώ συγγνώμη. Μόλις μου με ενημέρωσαν ότι πρώτου να ε, φύγουμε από το θέμα των απορριμμάτων, ε, να θέσω το ερώτημα του Βιτόριο Πρόντι. Στον κατάλογό σας είναι το σημείο 3. Ο Επίτροπος Ποτότσνικ έχει προσπαθήσει να, να απαντήσει πολύ σύντομα στην ερώτηση αυτή, αλλά δεν είναι ικανοποιητική αυτή. Στις 20 Ιανουαρίου είπε ότι ναι, η Κομισιόν θα πρέπει να κάνει κάποιες έρευνες. Μιλάμε για την ε, επανεξέταση της ε, παλιάς οδηγίας για τα απορρίμματα, για, τις, ε, για τα απορρίμματα από ε, τι γίνεται λοιπόν με το θέμα των πλαστικών ε, ε, συσκευασιών, ιδιαίτερα με τις σακούλες. Έχουμε, έχουμε προχωρήσει ένα βήμα όσον αφορά την συνείδηση των καταναλωτών, αλλά θα ήθελα να ξέρω εάν να ξέρω αν έχετε σημειώσει πρόοδο στο θέμα αυτό. Ε, ευχαριστώ πολύ. Ο Νίκος Χρυσόγελος. Παρακαλώ. Και μετά ο Ρίχαρτ Ζήπερ. Μήπως υπάρχει κάποιος που δεν τον είδα. Όχι από ό,τι βλέπω. Ε, για να μην φύγουμε από την συζήτηση που κάνουμε για την ε, την ιεράρχηση στη διαχείριση των αποβλήτων, ε, θα αναφερθώ στην ερώτηση 2 Ζήλ Evans, ε, που αφορά αν η Κομισιόν έχει πραγματικά πλήρη κατάλογο ποιες χώρες έχουν κάνει ήδη την ενσωμάτωση της οδηγίας, αλλά ήθελα και να υπενθυμίσω μια παλιότερη ερώτηση που είχε κάνει η κυρία Ρεμπέκα Χάρμ σε σχέση με την διαδικασία με τη Γερμανία. Ε, είχε απαντήσει η Κομισιόν σε σχετική ερώτηση τον Αύγουστο του 2011 ότι το σχέδιο για την νομοθεσία που είχε περάσει η Γερμανία δεν ήταν πολύ συμβατό ε, σε σχέση με την ιεράρχηση γιατί αντιμετώπιζε την καύση των απορριμμάτων ε, από, ένα, από μια τιμή και πάνω από 11.000 ε, κιλοτζάουλ ανά κιλό ως ισοδύναμο με την διαδικασία ανακύκλωσης. Και είχε παραδεχτεί η Κομισιόν ότι αυτό δεν είναι συμβατό με την ιεράρχηση της, που επιβάλλει το άρθρο 4 της οδηγίας, ζήτησε να υπάρξει αναθεώρηση του άρθρου, αλλά δεν έχουμε καμία κίνηση από την ε, πλευρά της Γερμανίας στο να αλλάξει ε, το άρθρο. Έχει κινηθεί κάποια διαδικασία από την Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ, ο Ρίχαρτ Τζέμπερ. Πρώτον, πρέπει να πω ότι η δική μου ερώτηση δεν απαντήθηκε σε καμία περίπτωση το επεξεργάζεστε. Ναι, πού, ποιο και τι κάνει. Έχω την αίσθηση ότι δεν απαντήθηκαν κι άλλες ερωτήσεις. Και ε, διαβάζω σήμερα στον τύπο ότι ο Επίτροπος Ταγιάννη ε, φτάνει σε προτάσεις για υπόγειες δράσεις μέχρι και 600 και 1000 μέτρα. Υπόγεια. Ε, εκείνη τα υπόγεια είδατα και ο Γιάνν Γκερμπράντι ε, μίλησε για μια Ευρώπη που να εξοικονομεί πόρους. Ε, ο μεγαλύτερος πόρος είναι τα σκουπίδια. 400.000 ε, θέσεις απασχόλησης, μείωση των ρήπων αντίστοιχη με 47.000, πόσα είπατε, δεν θυμάμαι, αυτοκίνητα. Και ο Επίτροπος Φωτόσινγκ θα πρέπει να κάνει συγκεκριμένες προτάσεις. Ακριβώς στη Νότια Ιταλία είναι οξύτατο το πρόβλημα. Δεν πρόκειται πλέον για πόρους, αλλά πρόκειται για ανθρώπινες ζωές. Ραδιενεργά απόβλητα στην Ήπεθρο και παράνομο εμπόριο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαζεύει κυριολεκτικά όλα αυτά τα χρόνια και δεν κάνει τίποτα. Και να έρθει ο Ορμόδιος Επίτροπος και να μας πει παρακαλώ τι γίνεται που ε, δεν έχουν εκκινήσει ε, προσφυγές επί παραβάσεις, τα περιφερειακά ταμεία ε, αδρανούν και περιμένουν δισεκατομμύρια. και Κοιτάξτε, δεν ήρθαμε εδώ για να το συζητήσουμε να πιούμε ένα καφεδάκι. Θέλουμε να μας πούν συγκεκριμένα πράγματα. Ευχαριστώ, Ρίχα Τσέπερ Δεν θέλει άλλο συνάδελφο το λόγο από ό,τι βλέπω. Ωραία. Να δώσουμε το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παρακαλώ να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις τώρα και να καλέσουμε και τον αρμόδιο επίτροπο, νομίζω το ακούσατε. Ε, είναι στα ζητήματα που πρέπει να διεκπαιρεώσουμε εμείς ως Επιτροπή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει το λόγο. Παρακαλώ. Thank you. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ ζητώ συγγνώμη και πάλι προς τον κύριο Άντερ που δεν απάντησα ε, για τις μεταφορές αποβλήτων. Είναι γνωστή η θέση μας Ανησυχούμε πραγματικά για την αποτελεσματικότητα των ελέγχων, ε, της αποστολής αποβλήτων και της κυκλοφορίας του στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορεί η μελέτη μας να οδηγήσει σε νομοθετική πρόταση. Δυστυχώς όμως, αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σας απαντήσω, δεν μπορώ να σας δώσω περισσότερες λεπτομέρειες. Άλλο θέμα είναι η εξέλιξη της παραγωγής αποβλήτων, για να τη χαρακτηρίσουμε έτσι. Σας είπα προηγουμένως ότι η Eurostat εκπονεί τώρα πιο πρόσφατες στατιστικές, οι οποίες θα αντανακλούν την κατάσταση για το 2010. Από ό,τι φαίνεται, ο όγκος των αποβλήτων που παράγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση μειώθηκε αισθητά από το 2009 μέχρι το 2010. Ισχύει αυτό. Δεν έχουμε όμως στοιχεία για να εντοπίσουμε ακριβώς την αιτία αυτής της σημαντικής μείωσης. Από ό,τι φαίνεται, μπορεί να έχει παίξει ρόλο βεβαίως η οικονομική κρίση, αλλά αυτό που έχει σημασία να γνωρίζουμε είναι ότι ε, σύμφωνα με την οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα, τα κράτη-μέλη είναι υποχρεωμένα να εγκρίνουν μέχρι το τέλος του 2013 ειδικά σχέδια για τη διαχείριση ε, των αποβλήτων. Και κατά τον ίδιο τρόπο τα προγράμματα αυτά θα πρέπει να είναι βασικό στόχος, το βασικό μέσο για να μειωθεί η παραγωγή αποβλήτων, ο όγκος τους δηλαδή. Προετοιμάζουμε πάλι κατευθυντήρες γραμμές για την πρόληψη παραγωγής αποβλήτων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το εγχείρημα, γιατί σε τελική ανάλυση ο καλύτερος ε, τρόπος είναι η αποφυγή της παραγωγής στην ιεράρχηση. Δεν το ξέχασα αυτό που ρωτήσατε. Ε, την ερώτηση του κυρίου Πρόντι. Αλλά φοβούμαι ότι δεν μπορώ να σας δώσω οριστική απάντηση σήμερα. Το επεξεργαζόμαστε. Αυτό το θέμα για τις πλαστικές ε, σακούλες Είναι θέμα του Επιτρόπου Ποτότσνικ. Της μιας ω πλαστικέ σακούλες είναι βασική προτεραιότητα του κυρίου Ποτότσνικ, αλλά είναι πολύ δύσκολο να πούμε το χρονικό ορίζοντα στον οποίο θα έρθει νομοθετική πρόταση. Το θέμα της βιοδιαθεσιμότητας θα ε, συμπεριλαμβάνεται και σε αυτή την νομοθετική πρόταση, αλλά είναι πολύ ευρύτερο θέμα. Έχει να κάνει με όλα τα πλαστικά και αυτό που θα κάνουμε εμείς μάλλον είναι να αρχίσουμε μια διαδικασία ε, προβληματισμού και περισυλλογής για τη βιοδιαθεσιμότητα με ένα χωριστό νομοθέτημα για τα πλαστικά απόβλητα. Ε, είναι και αυτό στο στάδιο της επεξεργασίας της υπηρεσίας μας τώρα. έγινε μια ερώτηση για την ιεράρχηση των αποβλήτων στη Γερμανία. Αυτό συνδέεται και με την ερώτηση της κυρίας Εύανς που αναφέρατε. Βεβαίως, Έχουμε πρόβλημα με την ερμηνεία που δίδεται ε, κατά τη μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο. Ήρθαμε σε επαφή με τις γερμανικές ε, αρμόδιες αρχές. Εξ όσων γνωρίζουμε, η ε, νομοθεσία δεν έχει ακόμα εγκριθεί στη Γερμανία για την εφαρμογή της οδηγίας αυτής. Δεν ξέρω εάν το κείμενο θα εγκριθεί από τη Γερμανική Βουλή με τρόπο που να εισαγάγει αλλαγές για το συγκεκριμένο ζήτημα, αλλά σίγουρα αν υπάρχουν προβλήματα... Στην ιεράρχηση των αποβλήτων στο γερμανικό δίκαιο θα το ε, κοιτάξουμε και αν χρειαστεί θα προσφύγουμε επί παραβάση, παραβιάση της νομοθεσίας. Σε ό,τι αφορά την τελευταία ερώτηση που έκανε ο κύριος Ζέμπερ, δεν ξέρω αν ήταν ερώτηση ή σχόλιο, δήλωση. Πάντως, πρέπει να σας πω ότι ασχολούμαστε πάρα πολύ σοβαρά με όλα αυτά τα θέματα που αφορούν την εφαρμογή ε, της νομοθεσίας περί αποβλήτων και αφιερώνουμε πάρα πολύ χρόνο αλλά και πόρους σε αυτή την προσπάθεια για να χειριστούμε ορισμένε περιπτώσει που είναι πραγματικά άκρο σημαντικέ. Και στην καμπανία, την κρίση που αναφερθήκατε ειδικά για την περίπτωση της Ιταλίας, κύριε Σέβε, να είστε βέβαιος ότι μας απασχολεί και είναι πολύ καλό παράδειγμα. Ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Δεν είναι η τελευταία φορά που θα συζητήσουμε αυτό το θέμα. Θα το δούμε και με τον αρμόδιο επίτροπο σε εκτενή συζήτηση με την ησυχία μας με τον απαραίτητο χρόνο. Σας ευχαριστώ καταρχάς. Ε, και ερχόμαστε στο σημείο 21 τώρα. Εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας για το Περιβάλλον. Παραδοσιακό θέμα στην Επιτροπή Περιβάλλοντος έχουμε 4-5 φορές το χρόνο την ευκαιρία να υποβάλουμε ερωτήσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έχω αρκετές ερωτήσεις. Ο Καρλ Χάιτς Φλόρενς έκανε την ερώτησή του, την έστειλε, δεν ξέρω. Θέλει και προφορικά. Dann gehen wir zwei. Jill Evans ist beantwortet. Οι ε, δύο της κύρια Εύαν έχει απαντηθεί, Βιτόριο Πρόντι επίσης. Τέσσερα, εφαρμογή τη περιβαλλοντικής νομοθεσίας της κυρίας Δελάγκε, η οποία απουσιάζει. Την εκπροσωπεί κανεί. Ο κύριος Ζίμπερ, ο κύριος Φλόρεντ. Η πρώτη μου ερώτηση για τα απόβλητα ε, απαντήθηκε, αλλά για το Ρίτς δεν μου απάντησε. Θα ήθελα να μου απαντήσει στην άλλη μου ερώτηση για το Ρίτς, που είναι η άλλη μου ερώτηση. Κυρία Χάση, παρακαλώ. Ε, Εξαιτία τη οικονομική κρίση, φαίνεται ότι σε ορισμένε τουλάχιστον χώρε υπάρχει μία τάση να μειωθεί η περιβαλλοντική προστασία και να επιστρέψουμε σε αντιλήψεις για την ε, ανάπτυξη που είναι προηγούμενων δεκαετιών. Και αυτή είναι μια περίπτωση που τη διαπιστώνουμε στην Ελλάδα. Υπάρχει η πρόθεση μια σειρά νομοθετικών ρυθμίσεων που φαίνεται ότι ε, προσπαθούν να παρακάμψουν την περιβαλλοντική προστασία. Υπάρχει η πρόθεση διαδικασιών όπως ονομάζονται fast track ε, και άλλων νομοθεσιών που φαίνεται ότι ε, για να διευκολυνθεί η πρόθεση επενδύσεων δεν θα εφαρμοστεί όπως θα έπρεπε η περιβαλλοντική νομοθεσία. Υπάρχουν ε, ρυθμίσεις που αφορούν την ε, νομο, τη μαζική νομοποίηση αυθερέτων κτηρίων για λόγους πρακτικούς και φοβάμαι ότι υπάρχουν και ορισμένες πιέσεις και από την ίδια την Επιτροπή για να ε, παρακαμφθεί η αυστηρή εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Ενώ ε, αντίθετα από ό,τι έχουμε στήσει πολλές φορές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και φαίνεται σε πολλές ευρωπαϊκές πολιτικές, η προστασία του περιβάλλοντος είναι και ένα εργαλείο για να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας και να προωθηθούν βιώσιμες μορφές οικονομικής δραστηριότητας. Δεν πρέπει να επιστρέψουμε σε μια αντίληψη της δεκαετίας του 50 του 60 που η ανάπτυξη θα καταστρέφει το περιβάλλον και θα ερχόμαστε εκ των υστέρων να πληρώνουμε μεγάλο κόστος για την αποκατάστασή του. Έχει η Κομισιόν ασχοληθεί με αυτό το θέμα ειδικά στις χώρες που αντιμετωπίζουν σοβαρή δημοσιονομική κρίση τώρα. Ευχαριστώ. Η Γιούτα Χάουκ, για την ερώτηση παριθμών 6. Μα την ερώτηση αυτή ουσιαστικά τη θέσαμε όλοι μαζί από κοινού το ψήφισμά μας για το προϋπολογισμό του 2012. Θέλουμε να μάθουμε εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ουσιαστικά και αληθινά είναι σε θέση από πλευράς προσωπικού να υποστηρίξει όλες τις διαδικασίες που χρειάζονται για τους ελέγχους τα κράτη-μέλη. Είναι σε θέση από πλευράς ανθρωπίνων πόρων, καν. Και το δεύτερο, θα παρακαλούσαμε να έχουμε μια τράπεζα δεδομένων για να μπορούμε και μόνοι μας να ψάχνουμε, να κοιτάμε τα δεδομένα αυτά για το πώς εφαρμόζονται τα νομοθετήματα και ποιες είναι οι ελλείψεις και πού χωλαίνει η κατάσταση. Γνωρίζουμε όλοι ότι η δημόσια πίεση μπορεί καμιά φορά να βοηθήσει και πάρα πολύ στην υλοποίηση ε, της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ιδιαίτερα στα κράτη-μέλη που ε, καυχόνται ότι είναι συνεπέστατα. Δεν ξέρω ποιος μπορεί να τα απαντήσει, ίσως αυτός που δεν με ακούει αυτή τη στιγμή. Εκτός αν καταλαβαίνει και γερμανικά, δεν το αποκλείω. Ε, θα δούμε τι έχει να πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κάρλος Λούτερ επόμενος και σαν του χάσει για το ρίτσο κύριος Χρυσόγελος και πάλι παρακαλώ. Η εφαρμογή της ε, οδηγίας ριτς είναι πάρα πολύ σημαντική, αλλά από τα στοιχεία που έχουμε φαίνεται ότι, έχει, ότι υπάρχει μεγάλη αδυναμία ή και αποτυχία στην, ε, στα πρώτα στάδια εφαρμογή. Ε, θα έπρεπε να εξεταστούν περίπου 20.000 φάκελοι. Ε, μάλλον από τους 20.000 φάκελους θα έπρεπε να εξεταστεί ένα 5% περίπου 1.000 φάκελοι. Αλλά τα στοιχεία δείχνουν ότι το 2009 είχαμε περίπου το 50% αυτών που εξετάστηκαν, που ήταν πολύ λίγοι φάκελοι, 30 μάλλον, το 50% δεν είχαν επαρκή στοιχεία. Το 2010 η ποιότητα ήταν ανεπαρκής για το 66% των φακέλων, δηλαδή περίπου στους 60% το 66%, και το 2011 σε 146 περιπτώσεις φάνηκε ότι είναι ανεπαρκής η φάκελη για το 90% των, των ε, περιπτώσεων. Εδώ δεν βλέπουμε καν βελτίωση που θα περίμενε κανείς να υπάρχει από χρόνο σε χρόνο, αλλά μια πλήρη αποτυχία στην, ε, στο πρώτο στάδιο την αξιολόγηση. Επίσης, ε, δεν έχουμε πρωτοβουλίες ε, από την Κομισιόν στο θέμα της, του restriction. Δεν υπάρχει καμία πρόταση από την Κομισιόν, δεν υπάρχει καμία ενέργεια μέχρι τώρα. και για την περίπτωση για το τη λίστα της, το candidate list ε, μέχρι τώρα έχουμε μόνο 74 ε, ουσίες από σύνολο 136. Ε, μήπως πρέπει να κάνει κάτι η Κομισιόν για να επιταχύνει τις διαδικασίες και να προχωρήσει μια σημαντική ε, οδηγία όπως είναι αυτή του Ρίτσα αλλά που δεν φαίνεται ότι έχουμε από τα πρώτα στάδια μια αποτελεσματική παρέμβαση. Ευχαριστώ πολύ κύριε Χρυσόγγελε ο κύριος ε, Φλόρεντς επίσης ερώτηση έχει βγει αυτή τη στιγμή. Η Μισελ Ριβαζή και πάλι ο κύριος Χρυσόγελος για το Ρίτς. Okay, δεν θέλει κανείς να ρωτήσει τίποτα άλλο. Τότε θα δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να απαντήσει στις ερωτήσεις που της έγιναν. Um, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είμαι από την, νομική, την υπηρεσία περιβάλλοντος και με νομικά ζητήματα. Θα εξετάσω την 5-6 και ένα κομμάτι της 4, της 4 και συνεργούν τα απαντήσεις το ερώτημα σχετικά με τη ορίτσου. Το ζήτημα της κυρίας Χάση, του που υπέβαλε ο κύριος Χρυσόγελος, σχετικά με τις επιπτώσεις χρηματοπιστωτικής κρίσης ε, στην εφαρμογή της ε, περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Μπορούμε να πούμε δύο πράγματα εδώ. Βλέπουμε ότι υπάρχει έλλειψη χρημάτων και δεύτερον οι αλλαγές ε, στην εθνική νομοθεσία προκειμένου να μπορούν να γίνονται κάποια πράγματα με χαμηλότερο κόστος. Τώρα, για τη χρηματοδότηση δεν έχουμε κάποιο ιδιαίτερο εποπτικό σύστημα για να ελέγχουμε κατά πόσον αυτά τα χρήματα πηγαίνουν στην προσφύρη περιβάλλοντος. Έχουμε κάποια στοιχεία που μας επιτρέπουν να δούμε κατά πόσον δεν ε, χορηγείται ε, ικανή προστασία στο Natura, σύμφωνα με το Natura 2000. Αν λάβουμε αυτές τις προφορίες, τότε μπορούμε να ελέγξουμε μέσω παραπώνων ε, πώς έχει η κατάσταση. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε. Και αυτό αναφέρθηκε και νωρίτερα, ότι υπάρχει ένα σημαντικό με συμμετοχή χρηματοδότηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το 2011 η Κομισιόν υιοθέτησε μια ανακοίνωση για την περιφερειακή πολιτική που συμβάλλει στην βιώσιμη ανάπτυξη στην Ευρώπη για το 2020 και ε, δήλωσε ότι θα πρέπει να χρησιμοποιούνται να χρησιμοποιείται ε, κοινωνική χρηματοδότηση για, τις, ε, για την πρόοδο σε αυτούς τους τομείς έχουμε κάνει εμεί ω ε, Γενική Διεύθυνση Περιφερειακή έκθεση και συχνά ε, παραδείσαμε ότι χρήματα δεν ε, δαπανώνται και μία από τις χώρες είναι η Ελλάδα. Έχουμε 66 περιπτώσεις προσφυγής κατά της Ελλάδος λόγω χιτά. το ποσοστό απορρόφησης της Ελλάδας είναι 80%. Τα χρήματα υπάρχουν, αλλά δεν χρησιμοποιούνται, δεν απορροφώνται. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί η task force που έχει συσταθεί για να βοηθηθούν οι ελληνικές αρχές να χρησιμοποιήσουν περισσότερα κοινωνικά κονδύλια. Υπάρχουν λοιπόν διαθέσιμα χρήματα, αλλά συχνά λόγω προβλημάτων που έχει η κυβέρνηση δεν χρησιμοποιούνται, δεν απορροφώνται αυτά τα ποσά. στην Σόφια παραδείγματος χάρη όπως υπήρχαν χιτά παρόν με αυτούς της ε, καμπανίας και μπορούν να χορηγηθούν μέχρι 180 εκατομμύρια ευρώ για να βελτιωθεί το σύστημα. Βλέπετε λοιπόν ότι πλευρά χρηματοδότηση, εντάξει, είναι γεγονό ότι έχουμε κάποια παραδείγματα περικοπών, αλλά Προσπαθούμε να πείσουμε τα κρατη μέλη να χρησιμοποιήσουν περισσότερο τα κονδύλια που τους χορηγούνται ε, στην περίπτωση της Ελλάδας ε, δεν ε, συμβαίνει κάτι τέτοιο δημιουργούμε μια task force και προσπαθούμε να τους βοηθήσουμε αυτά σε ό,τι φορά το χρηματοδοτικό ζήτημα τώρα για τις νομικές αλλαγές στην Ελλάδα έχουμε μια κατάσταση στην οποία παρακολουθούμε τους σύνεγγυ. Ε, βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποιες μεταρρυθμίσεις που αφορούν το habitat και να ξέρετε ότι παρακολουθούμε στενά τα, τι συμβαίνει στην Ηνωμένο γιατί σχετικά με το ζήτημα αυτό. Ε, ο αρμόδιος υπουργό στη Βρετανία δήλωσε ότι ο φορέας ο είχε αντιμετωπίσει κάποια προβλήματα λοιπόν να είστε βέβαιοι ότι παρακολουθούμε πολύ στενά τις εξελίξεις ε, και η Κομισιόν θέλει να στείλει ένα θετικό μήνυμα. Δηλαδή ότι το προσφύγιο περιβάλλοντος ε, δεν ε, αντιτίθεται, δεν λογοθοκοπείται θα λέγαμε με τις εξοικονομήσεις και τις οικονομίες που θέλουν να γίνουν Αυτά σε ό,τι φορά την ερώτηση 5, ερώτηση 6 της κυρίας Χάουγκ. Ως επικεφαλής ε, της μονάδας ε, για τις παραβάσεις ε, προσπαθώ να λαμβάνω περισσότερα κονδύλια από το κοινοβούλιο αστευόμενος το λέω αυτό τώρα. Δεν έχουμε επανέλθει στο θέμα των χιλίων ε, περιπτώσεων ε, και μπορέσαμε να ελέγξουμε το 20% των περιπτώσεων σε φορά τις περιφερειακές στο 35% και έχουμε στα 260 περιπτώσεις έχουμε ε, ολοκλήρωση της, τα 2 τρίτα για τις 60 ε, περιπτώσεις που αναφέρατε κυρία Χάουγκου έχουμε Τέσσερι ε, περιπτώσει που βρίσκονται ενώπιον δικαστηρίων, Βέλγιο, Λουξεμβούργο και Ιρλανδία για το για ζήτημα πολεοδομικά, χωροταξίας. Τώρα η Συνδίκη Λισαβόνα μας επιτρέπει να ε, προσφύγουμε κατά των κρατών εάν ε, δεν μεταφέρουν την ε, οδηγία. Υπήρξαν δύο-τρει περιπτώσει με την Πολωνία και όπως ανέφερε και προηγούμενα ο συνάδελφος έχουμε 7 περιπτώσεις που θα εξεταστούν σύντομα για το ζήτημα της μεταφοράς της οδηγίας περί αποβλήτων. Αυτά σε αφορά τη δράση κατά των παραβάσεων. Έχουμε πολλά άτομα που ασχολούνται και δεν είναι μόνο δικηγόροι που ασχολούνται με το ζήτημα τη παράβαση, όπω στην περίπτωση τη καμπανία δεν είναι από δικηγόρους αλλά από την ομάδα του Βούλιο, σε άλλες περιπτώσεις χρησιμοποιούμε τεχνικούς. Έχουμε 500 εκατομμύρια κατοίκους. Όπω καταλαβαίνετε εμεί που ασχοληθούμε με ένα πολύ μικρό κομμάτι των ε, παραβάσεων. Πώς θα γίνει λοιπόν το άλμα για μια καλύτερη εφαρμογή. Ξέρετε πως η εφαρμογή αποτελεί προτεραιότητα για τον Επίτροπο. Το έχει αναφέρει επανειλημμένα. Ευτυχώς ε, την προσεχή εβδομάδα η Κομισιόν θα υιοθετήσει μια ανακοίνωση για, τον, ε, για την περιβαλλοντική νομοθεσία και νομίζω ότι εσείς είστε αυτοί οι οποίοι κρατάτε το λάβαρο Και ε, τώρα επανέρχομαι στην ερώτηση της κυρίας Χάουγκ. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η γνώση και η διάδοση αυτής. Δεύτερον, ε, ανταπόκριση και επιβολή. Συμφωνώ με την κυρία Χάουγκ ότι η ενεργός ε, ε πρόθεση της ενημέρωσης είναι κάτι το οποίο μπορεί να ασκήσει πίεση τα κρατημέλη γι' αυτό στην ανακοίνωση. Θα δείτε, εάν φυσικά εγκριθεί όπως έχει προγραμματιστεί, από το Σώμα των Επιτρόπων, τα ζητάει από τα κράτη-μέλη να θέσουν περισσότερες πληροφορίες στο διαδίκτυο, όπως κάναμε και για τα λουτρά και τα ύδατα αλουωμένων, αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο και ε, κάτι ακόμα είναι να έχουμε IPPC, τους ΧΙΤΑ, τους εξοδετωμένους να αναρτηθούν στο διαδίκτυο. Το παράδειγμα λοιπόν της ε, οδηγίας για τα ύδατα λουμένων ε, είναι πάντα παρόν θα λέγαμε και μας βοήθησε πάρα πολύ στην εφαρμογή. Θέλουμε να βάλουμε περισσότερες προφορίες στην ε, διαδίκτυο προκειμένου οι πολίτες να μπορούν να ενημερωθούν και να ασκήσουν αν θέλετε πίεση μέσω ελέγχων στο κράτος τους. Και τώρα παίρνουμε στο θέμα των ε, χιτά, όταν έχουμε καταλόγους ε, με, τις, ε, με τους χιτά, τότε μπορείτε να ξεχωρίσετε τους νόμιμους από τους παράνομους. Επίσης κάνουμε ελέγχους για διαχείριση απορριμμάτων. Υπάρχουν οι εθνικοί μηχανισμοί προσφυγής. Θέλουμε να υπάρχει καλύτερη πρόσβαση στην δικαιοσύνη. και συμφωνίες τελικής σχέσης με τα κράτη-μέλη και να ζητήσουμε τα κράτη-μέλη να εστιάσουν τη χρηματοδότηση προγραμμάτων τα οποία είναι υποφελή για το περιβάλλον. Θα ήθελα να ολοκληρώσω με το ζήτημα της διαφάνειας ε, πλευράς Κομισιόν. Επ' αυτού η θέση της Κομισιόν είναι σαφής η βάση δεδομένων που χρησιμοποιείται για την ε, διαχείριση περιπτώσεων παράβασης δεν είναι δημόσιες. Υπάρχουν ε, πάντα δύο εμπλεκόμενοι. Η διαδικασία όμως ε, προστατεύεται από διότι δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στην βάση δεδομένων. Αυτό είναι Τώρα, σε ό,τι φορά την πληροφόρηση για την προαγωγή της ε, ενημέρωσης, τότε αυτό είναι δυνατόν. Αυτό καλύψαμε το 5 και το 6, να περάσουμε τώρα στο 6, έχουμε reach. Για το REACH σας παρακαλώ δεν απαντήσατε. Σας ευχαριστώ ε, για την εκτενή σας αναφορά. Ε, πολύ συγκεκριμένα όλα αυτά που μας είπατε, αλλά για το Ρίτσελμα να μας πείτε τώρα. Thank you very much, Mr. Chairman. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Λέγομαι Πιόν Χάνσεν από την ε, Μονάδα ε, Χημικών στη Γενική Διεύθυνση ε, για το Περιβάλλον και θα απαντήσω στα τρία ερωτήματα που έχουν να κάνουν με το REACH από τους βουλευτές και χαίρομαι πολύ για τον διάλογο αυτόν. Οι τρεις ερωτήσεις ήταν ε, η μία για την αξιολόγηση, η άλλη για τους περιορισμούς και η τρίτη για την αδειοδότηση. Ε, και οι τρεις ερωτήσεις ε, ήταν, για να συνοψίσω, αν η ήταν ποια είναι η πρόοδος και η απάντηση είναι πράγματι ότι η απάντηση δεν είναι, η, η πρόοδος δεν είναι η επιθυμητή, μπορούν να γίνουν κάποια πράγματα, έχει σημειωθεί όμως και κάποια πρόοδος. Ε, να αναφερθώ όμως στον καθένα από τους τρεις τομείς και να απαντήσω. Να ξεκινήσω από την αξιολόγηση. Νομίζω ότι είναι σημαντικό, προτού να απαντήσω στην ίδια την ερώτηση, να αναφέρω ότι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών στο Ελσίνκι εφαρμόζει κριτήρια για να επιλέξει ουσίες ε, οι οποίες θα πρέπει να ελεγχθούν σχετικά με τη συμμόρφωσή τους. Αυτό σημαίνει ότι εξετάζεται ο φάκελος των ουσιών για να δουν αν ε, συμμορφώνονται με τις ε, απαιτήσει του REACH. Κατά την ανάπτυξη αυτών των κριτηρίων ψάχνουν φακέλους που είναι πιο πιθανό να μη συμμορφώνονται. Γι' αυτό σαφώς αν κοιτάξει κανείς μόνο τα νούμερα στην ιστοσελίδα ή στην ετήσια έκθεση της, ε, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών φαίνεται να υπάρχουν ε, περισσότεροι φάκελοι που δεν συμμορφώνονται από ό,τι μπορεί να υπάρχουν συνολικά ως ποσοστό. Αλλά το ποσοστό μη συμμόρφωσης είναι πράγματι υψηλό και γι' αυτό ανησυχεί και την Κομισιόν αν και θα έλεγα ότι αυτό δεν είναι τελείως αναπάντεχο δεδομένης της καινοτομίας ε, της διαδικασίας ε, καταχώρησης καθώς και λόγω της πολυπλοκότητας ε, των υποχρεώσεων του σχετικού βιομηχανικού τομέα. Η Κομισιόν εδώ και χρόνια ζητάει από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών να κοιτάξει να θεωρήσει την αξιολόγηση προτεραιότητα ε, γενικά, αλλά ειδικά την, ε, ε, τον έλεγχο της συμμόρφωσης των χημικών. Σίγουρα λοιπόν αυτό αποτελεί σημαντική προτεραιότητα για τον οργανισμό μας. Αυτή τη στιγμή κοιτάμε το υψηλό ποσοστό μη συμμόρφωσης, εξετάζουμε το ποσοστό αυτό για να δούμε μήπως υπάρχουν περισσότερα που μπορεί να κάνει η Κομισιόν. Και Σκοπεύουμε να αναφέρουμε τα αποτελέσματά μας και να υποβάλουμε και συστάσεις σχετικά με το τι θα πρέπει να κάνουν οι Κομισιόν και άλλοι φορεί ε, στα πλαίσια της αναθεώρησης ε, του ΡΙΤΣ που ε, σχεδιάζουμε να ολοκληρώσουμε σύμφωνα με την προθεσμία που υπάρχει στον κανονισμό ΡΙΤΣ μέχρι τον Ιούνιο δηλαδή φέτος σκοπεύουμε να ολοκληρώσουμε τις εργασίες αυτές. βλέπουμε λοιπόν, θεωρούμε, και εμείς ανησυχητικά τα νούμερα αυτά και τα εξετάζουμε στα πλαίσια της αναθεώρησης του ΡΙΤΣ. Όσον αφορά τους περιορισμούς και εδώ προτού να μπω ε, σε λεπτομέρειες σχετικά με την πρόοδο που έχουμε σημειώσει θα θέλαμε να επαναλάβουμε ότι υπάρχει σαφής δέσμευση από πλευράς της Κομισιόν να ε, επιδεχθούν οι στόχοι ε, του Ρίτσε να ε, έχουμε καλή προστασία της ανθρώπινης υγείας ε, του περιβάλλοντος, καλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, καθώς και προώθηση της ανταγωνιστικότητας το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή η Κομισιόν δεν έχει ζητήσει από τον ε, Οργανισμό Χημικών της Ευρώπης να ετοιμάσει ε, φακέλους ε, σύμφωνα με το παράρτημα 16 για νέες ουσίες, ουσίες που δεν βρίσκονταν υπό έλεγχο στο παρελθόν. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να βγάλουμε συμπεράσματα σχετικά με την εξέταση ουσιών που μπορεί να, ε, που πιθανότατα να αποτελούν κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Να σας πω όμως και κάποια πράγματα όσον αφορά την πρόοδο που έχουμε σημειώσει ε, τα τελευταία χρόνια. Καταρχήν, Σύμφωνα με τις απαιτήσει του κανονισμού ΡΙΤΣ έχουμε ε, επεξεργαστεί κάποια μεταβατικά μέτρα ε, που έχουν να κάνουν με τα, περι... περιοριστικά μέτρα και έχουμε υποβάλει προτάσεις σχετικά με τους περιορισμούς που πρέπει να υπάγονται στο ΡΙΤΣ ε, και αυτό αφορά ιδιαίτερα δύο ουσίες, την ακριλαμίδη που το συμπεριλήφθηκε στο σχετικό παράρτημα του Ρίτσε, καθώς και το κάδμιο. τον Νοέμβριο του 2009 η Κομισιόν ζήτησε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών να ετοιμάσει έναν φάκελο ε, για τα περιοριστικά μέτρα ε, σχετικά με τον υδράργυρο σε ε, συσκευές μετρήσεως. Αυτή τη στιγμή τελειοποιεί τον φάκελο αυτό, ώστε να μπορέσουμε εμείς κατόπιν να κοιτάξουμε πού έχουν εντοπιστεί οι κίνδυνοι. Επίσης, φέτος, σε συναρχή του χρόνου, εξετάστηκαν ε, ε, περιοριστικά μέτρα για ουσίες που έχουν θεωρηθεί καρκινογόνες ε, και τοξικές για την αναπαραγωγή και μεταλλαξιογόνες και επίσης έχουμε προσαρμόσει και το παράρτημα 7 ε, του ΡΙΤΣ για δύο ουσίες με βάση δουλειά που έγινε υπό την προηγούμενη νομοθετική θητεία. Ουσιαστικά η διαδικασία περιοριστικών μέτρων Μάλλον συνοψίζοντας θα έλεγα ότι η Κομισιόν επικεντρώνεται στην ολοκλήρωση της δουλειάς που δεν ε, είχε ολοκληρωθεί ή που χρειαζόταν επανεξέταση από την ε, προηγούμενη νομοθεσία και στον τομέα αυτόν έχει σημειωθεί αρκετή πρόοδος, όπως βλέπετε. Όσον αφορά τα περιοριστικά μέτρα, σημαντικό είναι να θυμόμαστε ότι όχι μόνο η Κομισιόν ότι δεν παίρνει μόνο η Κομισιόν ε, την πρωτοβουλία, ε, αλλά και τα κράτη-μέλη συμμερίζονται την ευθύνη αυτή της Κομισιόν να ε, ξεκινούν διαδικασίες για περιοριστικά μέτρα και να, κάνουν, να επιβάλλουν αντίστοιχη αίτηση στην, ε, στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών ε, όταν εντοπίσουν σχετι, πιθανό κίνδυνο. Αυτή τη στιγμή κοιτάμε και την εφαρμογή των παρόντων περιοριστικών μέτρων. Κάτι τέτοιο φαίνεται να ε, περιορίζει κάπως ε, τον ενθουσιασμό των κρατών μελών ε, να υποβάλουν νέες προτάσεις για περιορισμούς στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών. Ε, στο επόμενο θέμα να ε, αναφερθώ σε κάποιες προτάσεις ε, του κ. Ταγιάννη και του Επιτρόπου Ποτότσνικ που ήθελε να επιταχύνει τις διαδικασίες για ουσίες που προκαλούν ιδιαίτερη ανησυχία. Η συμφωνία που έγινε τον Μάιο του 2010 σύμφωνα με τη συμφωνία αυτή ε, είπαν ότι θα πρέπει να επιτευχθεί ένας στόχος 106 ε, ουσιών μέχρι το 2012 και συμφώνησαν επίσης ότι θα πρέπει όλες οι αυτή τη στιγμή γνωστές ε, ουσίες που πληρούν τα κριτήρια να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το 2020. Έχουν θέσει λοιπόν πολύ συγκεκριμένο στόχο σχετικά με το τι θέλουν ε, ο Επίτροπος και ο Αντιπρόεδρος ε, να επιτευχθεί. Αναγνωρίζοντας το ρόλο του οργανισμού ε, χημικών, οι Επίτροποι σε επιστολή προς τις μόνιμες αντιπροσωπείες, προς μόνιμους αντιπροσώπους, τόνισαν ότι βασίζονται στην συνεργασία των κρατών μελών για τον αντιμετωπισμό των ε, σχετικών ε, ουσιών, ε, ενώ ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών θα κάνει την υπόλοιπη δουλειά. Και πάλι βλέπουμε δηλαδή μοιρασμένη αρμοδιότητα. Έκτοτε έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος, για παράδειγμα, η Επιτροπή μαζί με τον Οργανισμό Χημικών και τα κράτη-μέλη έχουν ξεκινήσει εργασίες πάνω σε ένα κοινό πλαίσιο για τις ε, ουσίες ε, που προκαλούν ιδιαίτερη ανησυχία και θέλω να συμπεριληφθούν οι ουσίες αυτές ε, σε έναν κατάλογο υποψήφιων ουσιών. Επίσης εντοπίζονται οι απαραίτητοι φορείς για, την, για τις εργασίες αυτές. Υπάρχουν ουσίες που έχουν εντοπιστεί ως καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες και τοξικές για την αναπαραγωγή. Ε, ο, ο λέει ότι σε αυτό το σημείο πάντα θαυμάζω τους ε, διερμηνεί που ε, πρέπει να μεταφράσουν τους όρους αυτούς σε άλλες γλώσσες. Προσπαθούμε να αναπτύξουμε περισσότερο τις τις 57 ουσίες στην κατηγορία F. Ε, υπάρχουν τώρα οι δυνατότητες ε, δημιουργίας ε, συνεργειών μεταξύ κρατών μελών με εταιρικέ σχέσεις, οικοδόμηση γνώσης μεταξύ των σχετικών φορέων. Υπάρχουν δηλαδή συνεργασίες πάνω σε συγκεκριμένε ουσίες ή ομάδες ουσιών. Ως αποτέλεσμα υπάρχει αύξηση των αριθμών στον κατάλογο το, στον αριθμό των ουσιών στον κατάλογο των υποψήφιων ουσιών. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε φτάσει τον στόχο των 136 ακόμα. Αυτή τη στιγμή πιστεύουμε ότι θα πρέπει να ενθαρρύνουμε τα κράτη-μέλη να επιταχύνουν περαιτέρω τι εργασίε. Ωστόσο, πιστεύουμε επίση ότι είναι σημαντικό η Κομισιόν και ο Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών να επιδείξουμε την ε, δέσμευσή μα να πετύχουμε τον κοινό μα στόχο. Και γι' αυτό η Κομισιόν από τη δική τη πλευρά ήδη έχει ζητήσει από τον Οργανισμό Χημικών να ετοιμάσει φακέλους για 10 ουσίες και ζήτησε από την ΕΚΑ, από τον ε, Οργανισμό Χημικών, να ε, δηλώσει τι δυναμικό έχει στη διάθεσή του για να ε, διαπιστωθεί αν μπορεί να καλύψει περισσότερους φακέλους από αυτούς που ζητήθηκαν αρχικά. Ζητήσαμε από την ΕΚΑ να ετοιμάσει άλλες, άλλους 15 φακέλους φέτος. Τέλος, ασχολούμαστε και με το πώς μπορούμε να επιτύχουμε το στόχο του 2020. Όλα αυτά μαζί ελπίζουμε ότι θα μας ε, βοηθήσουν να αυξήσουμε τον αριθμό στον κατάλογο των χημικών. Καταλαβαίνω ότι αυτή ήταν μια μακροσχελής απάντηση ε, στις τρεις προφορικές ερωτήσεις. Ευχαριστώ μπορώ να επανέλθω και σε κάποιες ερωτήσεις που δεν ε, τέθηκαν, ε, τις οποίες όμως είχαμε την τύχη να λάβουμε ε, εκ των προτέρων. Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, ευχαριστώ πραγματικά εκτενέστατη η απάντησή σας στις ερωτήσεις μας. Ο Κρίς Δέβης έχει ζητήσει το λόγο, δεν ξέρω. Ο Καλ Σλούιτερ τι κάνει εδώ από που πήγαινε έρχεται μέσα στην αίθουσα. Θέλεις το λόγο Κάρλα. Όχι. Εγώ είμαι στην ακρόαση για την άκτα. Ε, θα μπορούσα να μα στείλει γραπτό στι απαντήσει για να τι διαβάσω μετά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα σα ήμουν ευγνώμων. Μάλιστα. Τα απάντησε ο άνθρωπος. Εντάξει. Θα σας διαβιβαστεί. Ο κύριο Κρι Ντέιβις έχει το λόγο. I was going to start by making the same point, Chairman. Και εγώ το ίδιο θα έλεγα, Πρόεδρε. Ε, είναι πολύτιμες αυτές οι συνεδριάσεις ε, αυτές τις συζητήσεις που κάνουμε για την εφαρμογή της νομοθεσίας και τις βάζουμε τελευταία ώρα στο τέλος της εβδομάδας των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών, εξού και η προσέλευση. Στο παρελθόν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορούσε να μας ε, δίνει γραπτό τις απαντήσεις. Ε, θα μπορούσατε να μας τις ξαναδώσετε γραπτός, γιατί έτσι θα μπορέσουν να υποφελθούν και οι άλλοι συνάδελφοι που απουσιάζουν τώρα. Για το REACH ήθελα να ρωτήσω κάτι συγκεκριμένο. Στην πρώτη ερώτηση, για τις ε, καταγραφές, τις καταχωρήσεις ε, των προβλημάτων. Αλλά είναι πολλές, αλλά δεν ξέρω αν είναι σημαντικές. Πώς αξιολογείται αυτό. Είναι λεπτομέρειες ή μήπως είναι κίνδυνος για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον. Ε, τι σημασία είναι, μπορείτε να απαντήσετε αυτό. Οι ελληματικές καταχωρήσεις. Ε, καλό είναι αυτό που είπατε και λέει ο Πρόεδρος για τη γραπτή απάντηση. Να το συζητήσουμε και στους συντονιστές. Τέτοια πράγματα καλό θα ήταν. Εμείς εφαρμόζουμε συνεχώς, ε, μάλλον ε, μαζικά αποφασίζουμε ε, νομοθεσία και δεν ξέρουμε τι συνέχεια δίδεται στην πράξη. Καλή η θεωρία, αλλά καλό είναι να την ελέγχουμε και την υλοποίηση και γραπτός να έχουμε τα στοιχεία. Παρακαλώ, κύριος Χρυσόγελος. Θα ήθελα να υπενθυμίσω και την προφορική ερώτηση ε, Μισελ Ριβάση για την ε, τέφρα που προέρχεται από την καύση των δημοτικών αποβλήτων. Ε, αν θέλετε να απαντήσετε γιατί ε, από ότι υπάρχει και η γνωμοδότηση επιβεβαίωση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων, πράγματι ε, εμπίπτει στο πλαίσιο του ΡΙΤΣ, αλλά δεν δηλώνεται ε, και η τέφρα αυτή προέρχεται από αποτέφρωση δημοτικών αποβλήτων, δεν καταχωρείται. Ε, και είναι πιθανό ότι ε, παράγεται ποσότητα πάνω από χιλίους τόνους τέφρας ετησίως σύμφωνα με τα στοιχεία, άρα αντιμετωπίζεται με παράνομο τρόπο έχει αντιμετωπίσει το θέμα η Κομισιόν, σχεδιάζει κάποιες ενέργειες πάνω στο θέμα. Ε, θα απαιτήσει να καταχωρείται η τέφρα που προέρχεται από την καύση των δημοτικών αποβλήτων και να μην χρησιμοποιείται ως ε, δευτερογενή πρώτη ύλη όπως σήμερα. Ευχαριστώ. Ολοκληρώθηκε ο γύρος των ερωτήσεων. Δεν θέλει κανείς άλλος συνάδελφος το λόγο. Δεν βλέπω άλλο συνάδελφο να ζητάει το λόγο. Ε, η ερώτηση του κυρίου Φλόρεντς, υπαριθμών 8. Θα παρακαλούσα επίσης να την απαντήσετε. Δεν βλέπω άλλους συναδέλφους, όχι απλώ να ζητούν το λόγο, δεν βλέπω άλλους συναδέλφους, τελεία. Παρόλο που έχουμε χρόνο μέχρι τις 6.30. Παρακαλώ να μας απαντήσετε τις υπόλοιπες ερωτήσεις και τη γραπτή του κυρίου Φλόρεντς, συμπαριθμόν 8. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Θα αρχίσω από ε, τις ε, ελληματικές καταχωρήσεις, που ρωτήσετε αν είναι λεπτομέρεια όχι και θα συνεχίσω με τα υπόλοιπα. Για τις ελληματικές καταχωρήσεις, αν είναι λεπτομέρειες αυτά που εμφανίζουν ως ελλείψεις. Προσπαθούμε να επικεντρωθούμε όχι τόσο πολύ στο θέμα της ποιότητας, αλλά στο θέμα της συμμόρφωσης. Δηλαδή είναι ελληματικές καταχωρήσεις ως προς την υποχρέωση συμμόρφωσης. Είναι μεγάλο το ποσοστό των φακέλων που δεν συμμορφώνονται, που δεν συμφορμώνονται με τις απαιτήσεις ενημέρωσης και πληροφόρησης. Δηλαδή, είναι ελλειπής η πληροφόρηση, η καταχώρηση, ο φάκελος. Αυτό είναι το πρόβλημα, ότι δεν δίδονται οι ε, σωστές πληροφορίες και αυτό ενδεχομένω μπορεί να έχει επίπτωση. Μπορεί, το τονίζω, στη διαχείριση του κινδύνου. Δεν σημαίνει ότι οφείλει. Αλλά το REACH έτσι οικοδομήθηκε γύρω από αυτή την έννοια της, ε, των ελάχιστων απαιτήσεων ενημέρωσης και πληροφόρησης και αυτό είναι παραβίαση και, ε, και μη συμμόρφωση με τις ελάχιστες αυτές τις πληροφορίες. Το θέμα λοιπόν δεν είναι η ελλειπής ποιότητα, αλλά οι ελληματικές καταχωρήσεις είναι έλλειψη πληροφόρησης που έπρεπε να δίδεται. Και αυτό προσπαθούμε να διορθώσουμε. Αυτά είναι τα ελλειπή στοιχεία. Δεν είναι ορθογραφικά λάθη, ας πούμε. Τώρα, ε, σχετικά με την τέφρα από την αποτέφρωση ε, των δημοτικών αποβλήτων. Ζητώ συγγνώμη, δεν μπορέσαμε σε μεγάλο βαθμό να το μελετήσουμε για να σας δώσουμε εμπεριστατωμένη απάντηση για λόγους έλλειψης χρόνου από τη στιγμή που κατατέθηκε η ερώτηση. Ζητώ συγγνώμη, ε, αλλά θα παραμείνω στην επιφάνεια, δεν θα μπω στο βάθος της απάντησης. Μπορώ να σας απαντήσω ότι θα χρειαστώ μεγαλύτερη μελέτη. Αυτό που διαπιστώσαμε Ε, στην ιστοσελίδα του JRC, του Ευρωπαϊκού Συστήματος ε, Πληροφόρησης για τις Ουσίες ε, που λειτουργεί, είδαμε ότι η τέφρα έχει κατοχωρηθεί εκεί. Από το 1993 ήταν ο κανονισμός, αν δείτε. Χρησιμοποιώ ε, την ορολογία του Ρίτς. Μιλώ για καταχωρήσεις. Τότε δεν το λέγαν καταχώρηση, αλλά καταλαβαίνετε τι εννοώ. Τότε είχε καταχωρηθεί λοιπόν από έναν Ολλανδικό όμιλο ήταν μία μοναδική ε, καταχώρηση και δεν ήταν ε, ευρία η γνώση γι' αυτό. Γνωρίζουμε όμως από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Οργανισμό Χημικών ΕΧΑ ότι δεν έχει ενταχθεί στο ΡΙΤΣ. Θα πρέπει να το δουν πρώτα οι συνάδελφοι αυτό στον Οργανισμό Χημικών Προϊόντων. Για ποιο λόγο υπάρχουν διαφορές, ενδεχομένω να υπάρχουν διαφορές ε, με τις πρακτικές του παρελθόντος και αν η συζήτηση με τους συναδέλφους εκεί του οργανισμού δείξουν ότι θα πρέπει να απευθυνθούμε στα κράτη-μέλη, θα το πράξουμε ως δεύτερο όμως βήμα. Πάντως θα το διερευνήσουμε με τους αρμόδιους συναδέλφους του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων. Επανέρχομαι τώρα στην ερώτηση 8 για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και το ΡΙΣ. Δεν θα επαναλάβω τις ερωτήσεις. Είναι πολλές εκείνες που αναφέρονται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στο χρονοδιάγραμμα αναθεώρησης αυτό καθ' αυτό. Θα διατρέξω λίγο τις απαντήσεις. Τι επιπτώσεις έχει το REACH ε, στις μικρομεσαίες τι παρατηρούμε. Θα το συμπεριλάβουμε στην αναθεώρηση του ΡΙΣ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει αυτό το καιρό θεματικές μελέτες για να δει πώς λειτουργεί το σύστημα. Σε δύο θεματικές μελέτες κοιτούν τον αντίκτυπο στις επιχειρήσεις και ε, μία ονομάζεται την, την βαφτίσαμε πάση περιπτώσει μελέτη αγοράς και καινοτομίας και επικεντρώνεται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και πάλι λοιπόν στην αναθεώρηση του REACH κοιτούμε τι επιπτώσεις έχει στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τα ευρήματα λοιπόν ε, μαζί ε, με τα όσα έχει αντλήσει από άλλες πηγές από την ομάδα επαφής της Διεύθυνσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που ήταν στις δόξες της ε, στα τέλη του 10 και στις αρχές του 11, όπως επίσης και ε, τη διάσκεψη για την καταχώρηση το Σεπτέμβριο του 2011 και το εργαστήρι του Δεκεμβρίου του 2011 για την γενοτομία και μια διάσκεψη που επίσης σήμερα διεξάγεται για την εφαρμογή του REACH Όλα αυτά λοιπόν είναι πηγές πληροφόρηση, πήραμε όλα τα στοιχεία και μαζί με τις τακτικές επαφές που έχουμε έτσι κι αλλιώς με τη βιομηχανία και τους ε, μεγάλους φορείς, έχουμε και το UE και PME που δεν προφέρεται <laughs> εν πάση περιπτώσει ως ε, αρχικά και αρκτικόλεξη, Έχουμε και ένα δίκτυο για τις μικρομεσαίες και μια εβδομάδα για τις μικρομεσαίες. Όλα αυτά τα στοιχεία τα συλλέγουμε λοιπόν και θα κάνουμε συστάσεις όπου χρειάζεται για να βοηθήσουμε ακόμα περισσότερο. για να δούμε πώς έχει η συμμόρφωση και τι σημαίνει αντίκτυπος. Σε ό,τι αφορά την αρχή, το σύστημα, μια ουσία, μια καταχώρηση, θυμάστε, όζορ λέγεται, στη διαδικασία συναπόφασης του Ριτς δεν ξέρω κατά πόσο αυτό προκαλεί μεγάλο ε, γραφειοκρατικό φόρτο, αυτό ρωτάτε. Ε, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων μας ενημερώνει και αν δείτε τα αποτελέσματα που γράφουν στην έκθεσή τους θα διαπιστώσετε ότι έχει επιτύχει αυτό το σύστημα. Είναι πραγματικά μεγάλο σουξέ. Το 90% των καταχωρήσεων έγιναν σε κοινέ λεγόμενες καταχωρήσει. Αυτή είναι η τεχνική ορολογία για το μια ουσία, μια καταχώρηση. Βεβαίω υπήρξαν κάποιες ε, δυσκολίες στην αρχή για τις κοινέ καταχωρήσει και το είδαμε στην ομάδα επαφή των διευθυντών, ε, αλλά τελικά έγιναν οι καταχωρήσει και οι φάκελοι ήρθαν κανονικά. ω μία ουσία μία καταχώρηση. Όπως σα είπα, το θέμα το παρακολουθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων και η ομάδα Επαφή των διευθυντών έχουμε εκπονήσει πολύ συγκεκριμένες λύσεις. Αναφέρει η βιομηχανία πώς λειτουργεί αυτό, όλα τα λέει στην ιστοσελίδα ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επόμενη ε, προθεσμία. Οι λύσεις για ένα κοινό πλαίσιο και πώς μπορούν να λειτουργήσουν θα έδιναν καλές ενδείξεις για το πώς γενικά λειτουργεί αυτό το σύστημα ανταλλαγή πληροφοριών για τις ουσίες, αν το σύστημα μία ουσία, μία καταχώρηση ε, λειτουργήσε, αν οι εταιρείε που καταχωρούν την ίδια ουσία το υιοθετούν. Πρέπει όμως να δημιουργήσουμε ε, οικονομία κλίμακος για να α, στείλουμε ε, στάνταρ ε, έγγραφα, έντυπα, κοινού κανόνε να υιοθετούν οι εταιρείε και τα λοιπά, για τα χρονοδιαγράμματα, για την ανταλλαγή πληροφοριών και ακόμα και με μέσα πληροφορικής να τις υποστηρίζουμε. Και η ομάδα επαφής των διευθυντών συνεχίζει τις εργασίες ακριβώς για αυτά τα θέματα. Αν μου επιτρέπετε τώρα έρχομαι στην τελευταία ερώτηση για την αναθεώρηση του REACH Μέχρι την 1η Ιουνίου του 2012 αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί αυτή η προσπάθεια. Εκεί προσανατολιζόμαστε. Θα πάρει τη μορφή ανακοίνωση προ το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο και θα υποστηριχθεί από ένα έγγραφο εργασία τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα γίνει δημόσιο διάλογο με τα δύο θεσμικά όργανα. Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτίθεται να έχει και δημόσια διαβούλευση με ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων και ενεχομένων. Προ το παρόν, ε, προγραμματίζουμε, σκοπεύουμε να κάνουμε μια διάσκεψη για τις συστάσεις στις 24 Σεπτεμβρίου αλλά έχουμε αρχίσει τις συζητήσεις από τώρα για να μπούμε ε, σε ένα πιο λεπτομερές πρόγραμμα μέχρι τότε. Σε αυτό το εργαστήριο, 24 Σεπτεμβρίου, έτσι κάπως ε, ενδεικτικά, πότε να περιμένετε την ανακοίνωση και την ολοκλήρωση της αναθεώρησης με τα απαραίτητα συνοδευτικά ε, έγγραφα. Ελπίζω να απάντησα στις ερωτήσεις σας, αλλιώς να μου το πείτε. Να προσπαθήσω ξανά. Αν έμεινε τίποτα αναπάντητο και αν επιθυμείτε, επανέλθω. Ευχαριστώ. Yeah. Κύριε Χάνζεν, σας ευχαριστώ πολύ και εσάς και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αναλυτική σας απάντηση και εκτενείς ερωτήσεις μας. Οι συνάδελφοι δεν ξέρω αν θέλουν να ρωτήσουν τίποτα άλλο. Οι δύο-τρεις συνάδελφοι που έχουν απομείνει ε, δεν έχουν ερωτήσεις, οπότε μπορούμε να ολοκληρώσουμε και αυτό το σημείο της μερισίας διάταξης. Θα το συζητήσουν οι συντονιστές το θέμα και την πρόταση του Chris Davis για το πώς μπορούμε να έχουμε και γραπτό απαντήσεις σας. Καλή πρόταση. Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ όλους όσοι συνεισφέρετε σε αυτή την προσπάθεια. Επόμενο θέμα και τελευταίο. Προσεχή συνεδρίαση. Η επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής μας λαμβάνει χώρα την 3η 20 Μαρτίου, 3 με 6.30. Τετάρτη 9 με 12.30 και το απόγευμα 3 με 6.30 και την 5η 22 Μαρτίου 9 με 12.30. Εντάξει κηρύσω το πέρα συνεδρίασης και σας εύχομαι καλό σας βράδυ. Και όσοι ταξιδεύετε προς τις πατρίδες σας, καλό ταξίδι. Σας ευχαριστώ πολύ.